Καλημέρα. Συνεχίζουμε τη συνεδρίασή μας. Σας καλωσορίζω. Παρακαλώ, καθίστε. Καθίστε, παρακαλώ. Συνεχίζουμε τις συζητήσει μας. Σας παρακολουθώ. Σημείο 14. Σας ε, καλωσορίζω. Σημείο 14. Πολιτική ακαιρεότητα της ε, Ευρωπαϊκής Επιτροπής και ειδικότερα ο διορισμός του Γενικού Γραμματέα της Ευρωπαϊκής Επιτροπή. Σα καλωσορίζω Καλωσορίζω και ε, τον Επίτροπο, τον κύριο Έντιγκερ, την ομάδα του. Σας ευχαριστώ ε, που απαντήσατε στις 134 ερωτήσεις που σας στείλαμε. Ήταν δύσκολο έργο αυτό ε, και για να απαντήσετε εσείς και για να τις διαβάσουμε εμείς τις απαντήσεις σας και λάβαμε τις απαντήσεις σας την Κυριακή στις 3 το πρωί μαζί με όλα τα υπόλοιπα έγγραφα. Βλέπετε εδώ μια ολόκληρη στίβα. Λάβαμε, σας ευχαριστούμε για όλα αυτά και για τη διαφάνεια βεβαίως που επιδείξατε, για να δούμε πού βρισκόμαστε ε, στην υπόθεση αυτή. Διαπιστώνουμε διάφορα στοιχεία. Αφενός υπήρξε μια έκπληξη στην, στην όλη διαδικασία. Τόσο, ως προς την, ε, τόσο για το Κολέγιο των Επιτρόπων όσο και για την δημοσιότητα. Τρία ε, ήταν μόλι τα άτομα που ήξεραν ότι πρόκειται να ακολουθεί αυτή η διαδικασία και κατά συνέπεια υπήρξε μόνο μία υποψηφιότητα ε, αρχικός. Όταν πλέον το μάθανε και άλλοι δύο, δεν υπήρξε κανείς που να ισχυριστεί ότι θα μπορούσε ενδεχομένως να έχει ακολουθεί και μια διαφορετική διαδικασία. Ξεκίνησε μια δημόσια συζήτηση μεγάλη και εκτενής. Δεύτερο θέμα, η όλη διαδικασία ε, που εγώ πιστεύω ότι ο διορισμός του Γενικού Γραμματέα ε, γενικά δεν είναι θέμα το οποίο ενδιαφέρει τη δημοσιότητα. Όμως το γεγονός ότι ο ίδιος ο, ε, ο, ο Γενικός Γραμματέας παρετείται σε μια συνεδρίαση και ο αναπληρωτής του ε, προάγεται ταυτόχρονα σχεδόν, αυτό είναι ένα θέμα που θέτει ερωτηματικά βεβαίως ε, αντίστοιχα ερωτηματικά έχουν ε, απασχολήσει και εμάς ε, και το Συμβούλιο βεβαίως. Γι' αυτό και σας καλέσαμε για να συζητήσουμε τα θέματα αυτά. Τρίτον, υπάρχει ε, μία ένταση μεταξύ ε, υπαλλήλων καριέρας και επιτρόπων. Ε, γιατί ε, κανονικά ε, υπάρχει μια διαδικασία. 20% λοιπόν του προσωπικού της Κομισιόν κανονικά δεν έχει περάσει από διαγωνισμό. Γνωρίζουμε όλοι ότι ένας τέτοιο διαγωνισμός για πρόσληψη στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι μια δύσκολη διαδικασία, την οποία δεν ακολουθούν όλοι. Βλέπουμε λοιπόν ότι υπάρχουν και άλλες διαδικασίε τι οποίες μπορεί να ακολουθήσει κανείς προκειμένου να προαχθεί ε, σε σχέση με αυτό που κάνουν οι περισσότεροι υπάλληλοι της Κομισιόν. Και βλέπουμε, για παράδειγμα, έναν τμήματάρχη, ο οποίος λόγω πολιτικής υποστήριξη έχει γίνει γενικός διευθυντή. Και λίγο, λίγους μήνες πριν από την λήξη της ε, της ε, θητείας της Κομισιόν βλέπουμε διάφορους αλεξιπτοτιστές ε, οι οποίοι αξιοποιούν ε, την, ε, το momentum, την ορμή που έχει δημιουργηθεί προκειμένου να αποκομίσουν προσωπικά ωφέλη. Βεβαίω αυτοί οι άνθρωποι στη συνέχεια καλούνται να πάρουν και πολιτικές αποφάσεις και πολιτική απόφαση σημαίνει ότι πρέπει κανείς να είναι ακέραιος και να ακολουθεί συγκεκριμένους κανόνες. Αυτή είναι και η θέση της Επιτροπής μας. Ο διορισμός του αναπληρωτή γενικού διευθυντή, γενικού γραμματέα ε, από εμάς επικρίθηκε γιατί ακριβώς θεωρούμε ότι είναι σημαντικό να εξασφαλίζονται ίσες ευκαιρίες για όλους τους υπαλλήλους. Και γι' αυτό το λόγο σας καλέσαμε να συζητήσουμε για την υπόθεση αυτού του νέου Γενικού Γραμματέα, έναν πολύ ικανό άνθρωπο βεβαίως, ο οποίος όμως ε, έχει ε, ακολουθήσει μια ε, εξαιρετικά γρήγορη προαγωγή και καριέρα. Δεν έχει κανείς βεβαίως αντίρρηση ότι ο άνθρωπος αυτός έχει ικανότητες, όμως δεν μπορούμε να καταλάβουμε, τουλάχιστον έτσι με μια πρώτη ματιά, για ποιο λόγο αυτός ο άνθρωπος θα έπρεπε να παρακάμψει και να ε, προσπεράσει ε, εκατοντάδες άλλους υπαλλήλους οι οποίοι θα μπορούσαν επίσης βεβαίως να έχουν θέση υποψηφιότητα και ε, είναι δεδομένο ότι έχουν και εκείνοι πολλές ικανότητες. Εγώ λοιπόν προσωπικά δεν έχω, δεν έχω καμία αμφιβολία για τις δεξιότητες και τις ικανότητες του νέου Γενικού Γραμματέα αλλά δεν είναι και αυτό το θέμα στην πραγματικότητα. Μιλούμε για την δημόσια συζήτηση η οποία έχει ξεκινήσει για αυτήν την υπόθεση και αυτή μας ανησυχεί. Γι' αυτό και θα ήθελα να σας καλέσω κύριε Επίτροπε να μας πείτε πώς θα αποκατασταθεί η ηρεμία ε, στην όλη συζήτηση. Κυρία Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, αγαπητοί ευρωβουλευτές, σας ευχαριστώ που μου δίνετε την ευκαιρία να συζητήσω μαζί σας, την αρμόδια δηλαδή επιτροπή, θέματα τα οποία έχουν βγει στην επιφάνεια της δημοσιότητας και να απαντήσω και στα ερωτήματα που μας αποστήλατε εσείς. Ε, θεωρώ ότι έπειτα από τη συζήτηση που έγινε στο Στρασβούργο, εδώ στο Κοινοβούλιο, ε, η σημερινή διαδικασία αποτελεί ε, μια χρήσιμη ε, συζήτηση που αφορά μια ευρύτερη συζήτηση και όχι μόνο τον διορισμό του συγκεκριμένου ε, Γενικού Γραμματέα. Θεωρώ λοιπόν με κάθε διαφάνεια θέλω ε, να απαντήσω στα θέματα που έχετε θέσει. Δεν θέλω να επαναλάβω αυτά που σας έχουμε ήδη απαντήσει μέσω των 134 απαντήσεων που σας αποστήλαμε, αλλά ε, θέλω να κάνουμε μια ευρύτερη συζήτηση. Είναι αλήθεια φυσικά ότι η θερινή ώρα ξεκίνησε στις 3 η ώρα το πρωί της Κυριακής. Και αυτό και ε, θέλω να πω κάτι ως προς τη διαδικασία που ακολουθήσαμε. Θεωρήσαμε ότι οι, οι απαντήσεις θα, οι, οι ερωτήσεις σας θα μας αποσταλούν τη Δευτέρα. Εντάξει, μια μέρα θα μπορούσαμε να, να ε, περιμένουμε. Μετά όμως είχαμε συνεδρίαση της Κομισιόν και μετά διήμερη σύνοδο κορυφής του ε, Συμβουλίου. Και έτσι ο πρόεδρος μου είπε ότι θέλει να αναλάβει και αυτός συνευθύνη σε σχέση με τις απαντήσεις που θα δώσουμε. Γι' αυτό και την ε, Τρίτη το βράδυ και την Τετάρτη η Γενική Διεύθυνση Ανθρώπινων Πόρων και στη συνέχεια η Νομική Υπηρεσία της Κομισιόν ε, εξέτασαν τις ερωτήσεις ε, και κατάρτισαν κάποια σχέδια απαντήσεων. Δεν ήταν εύκολη αυτή η διαδικασία. Ήταν δύσκολο το έργο αυτό, διότι η δομή του καταλόγου ε, των ερωτήσεων ήταν κάπως ε, θολή. Δηλαδή υπήρχαν κάποιες ερωτήσεις οι οποίες δίνανε ε, αφορούσαν το ίδιο θέμα, ε, επικαλύπτονταν κτλ. κτλ. Εντάξει, δεν θέλω να σας ε, κάνω φθηνή κριτική, αλλά ήταν δύσκολη αυτή η διαδικασία. Εγώ στη συνέχεια την Παρασκευή, αφού γύρισα από τη Σύνοδο Κορυφής, γύρισα στο γραφείο μου και είδα ε, ότι το επιτελείο μου είχε ήδη... Ε, ε, συντάξει κάποιες απαντήσεις. Το Σάββατο λοιπόν έγινε μια τελευταία εξέταση των απαντήσεων που θα σας δίναμε και μέχρι τη νύχτα ε, χρειάστηκε να δουλέψουμε συντακτικά επί της διατύπωσης και στη συνέχεια σας αποστήλαμε ε, την, τις απαντήσεις μας. Δεν έχει καμία σχέση λοιπόν με τη θερινή ώρα, αλλά ακριβώς θέλαμε να ακολουθήσουμε διεξοδική διαδικασία σε βάθος προκειμένου να μπορέσουμε να απαντήσουμε στα ουσιώδη θέματα ώστε εσείς την Κυριακή και τη Δευτέρα να μπορείτε να εξετάσετε τις ε, απαντήσεις μας για να προετοιμαστείτε καλύτερα και για τη σημερινή μας συζήτηση. Και νομίζω ότι με, ακολουθώντας αυτήν την ε, ε, διαδικασία τόσο η Επιτροπή Κοντ όσο και η Κομισιόν ε, δουλέψαμε διεξοδικά και όχι ερασιτεχνικά. Για μας λοιπόν υπάρχουν δύο ομάδες ερωτημάτων που έχουν ουσία. Πρώτον, αν ο διοριστής από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, νέος Γενικός Γραμματέας, έχει τις ουσιαστικές και προσωπικές ικανότητες και τα προσόντα στη βάση της ε, εκπαίδευσής του, της ε, επαγγελματικής του εμπειρίας, ε, της επαγγελματικής του πορείας, των ικανοτήτων του, της ευφυΐας του, αλλά και της ε, προσωπικής του ακαιρεότητας αν έχει λοιπόν τα προσόντα για να διοριστεί. Βεβαίως η άποψη, ε, καθένας μπορεί να έχει τη μία ή την άλλη άποψη. Εγώ όμως τον γνωρίζω από κοντά εδώ και 8 χρόνια και πιστεύω προσωπικά και το ίδιο πιστεύει και ο πρόεδρός μου αλλά και οι συνάδελφοί μου ότι έχει τις τεχνικές, επιστημονικές και προσωπικές ικανότητες και προσόντα προκειμένου να εκπληρώσει τα καθήκοντα του Γενικού Γραμματέα. Βεβαίω είμαι στη διάθεσή σας για να μου πείτε διαφορετική άποψη αν έχετε. Μπορούμε και να διαφωνήσουμε, αλλά η δική μου άποψη ε, είναι ε, σταθερή. Αν έχει και τις νομικές προϋποθέσεις προκειμένου να καταλάβει θέση ε, στο επίπεδο στο οποίο διορίστηκε. Ναι, η απάντηση είναι ναι. Και αυτό προκύπτει από τον ε, κανονισμό ε, του προσωπικού. Δεύτερον, δεύτερο ερώτημα. Αν η διαδικασία που ακολουθήθηκε ήταν νομικά σωστή. Μπορεί κανείς βεβαίως να εξετάσει το γράμμα ή και το πνεύμα των κανόνων. Εγώ είμαι νομικός και δεν είναι πάντοτε εύκολο να διακρίνει κανείς το γράμμα και το πνεύμα, διότι πρόκειται για ένα, για, για, ένα και το αυτό κείμενο, το οποίο το staff regulation, το, το, κανονισμός του προσωπικού, όπου ε, συνδυάζονται και το γράμμα και το πνεύμα. Και ακριβώς επειδή το ερώτημά σας, τα ερωτήματά σα αφορούν περισσότερο το γράμμα των κανόνων, οι απαντήσεις μας επικεντρώθηκαν στη νομική διάσταση στη νομική και τεχνική ε, διάσταση του θέματος ως προς το περιεχόμενο των κανόνων που από γράμματα και λέξεις συνιστούν κανόνες για την προαγωγή και το διορισμό στελεχών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Εξετάζοντας ξανά και ξανά λοιπόν το κείμενο, Είμαστε πεπισμένοι για, την, για τον νόμιμο χαρακτήρα τόσο της διαδικασίας που ακολουθήθηκε όσο και του αποτελέσματος στο οποίο καταλήξαμε. Σε κάποια ερωτήματά σας ε, κάνετε παραπομπή σε κάποια έγγραφα στα οποία ζητάτε πρόσβαση. Κάποια από αυτά δικαίως θεωρούμε εμείς προστατεύονται από τους κανόνες για την προστασία προσωπικών δεδομένων. Γι' αυτό και δεν είναι εύκολο να σας δώσουμε πρόσβαση. Και γνωρίζω ότι και εδώ στο Κοινοβούλιο θεωρείται πάρα πολύ σημαντικό θέμα την προστασία των προσωπικών δεδομένων. Το να είναι, είναι, είναι λοιπόν τουλάχιστον ε, περίεργο να ε, μιλά το Κοινοβούλιο ε, Διαρκώ για την προστασία των προσωπικών δεδομένων και στη συνέχεια σε μια τέτοια περίπτωση να ζητάτε προσωπικές, προσωπικά δεδομένα ενός ανθρώπου που δεν μπορούν να παραβιαστούν. Παρ' όλα αυτά προσερχόμαστε εδώ στη συζήτηση ε, με την Επιτροπή σας προκειμένου με τις απαραίτητες ε, προϋποθέσεις να εξασφαλίσουμε την πρόσβασή σας στα προσωπικά δεδομένα του κυρίου Σελμαϊρ. Και το λέω αυτό συνειδητά προκειμένου να ε, ε, απαντήσω σε, σε πιθανές αμφιβολίες που μπορεί να εκφραστούν. Όχι για να υπονομεύσω το ισχύον δίκαιο. Αυτό θα έθετε σε κίνδυνο την ε, συνεργασία μας και δεν θα ήταν ούτε στο, στο συμφέρον του Κοινοβουλίου, ούτε της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ούτε και της εικόνας μας προς τα έξω, προς την δημοσιότητα, αλλά ούτε και προς το συμφέρον του ίδιου του Μάρτιν Σέλμαερ, ο οποίος ε, βεβαίως θα έπρεπε ε, επίσης να ε, ε, έχει, να, να έχουμε τη σύμφωνη γνώμη του για ό,τι κάνουμε με τα δικά του προσωπικά δεδομένα. Δεν πρέπει λοιπόν να δημιουργηθεί ένα αρνητικό προηγούμενο για το μέλλον. Θέλουμε να κάνουμε ό,τι περνά από το χέρι μας ώστε ε, εκπρόσωποι της Επιτροπής σας σε ε, ασφαλισμένη αίθουσα να έχετε εσείς και τα, τα μέλη της Επιτροπής σας πρόσβαση σε αυτά τα έγγραφα στις απαντήσεις μας ε, που δώσαμε ε, το Μάρτιο στο Στρασβούργο είχα μιλήσει για ένα πακέτο ε, κανόνων και εγγράφων. Κάποιοι από, αυτά, κάποιοι από αυτούς τους κανόνες έχουν ήδη εφαρμοστεί, κάποιοι βρίσκονται στο στάδιο της εφαρμογής τους. Έχει ξεκινήσει δηλαδή η προετοιμασία. Και έτσι ε, έχει ξεκινήσει ήδη μια διαδικασία για δύο αναπληρωτές γενικούς γραμματείς και ε, για ε, νέους γενικούς διευθυντής, συγκεκριμένα στην DG Εμπορίου και η ολοκλήρωση αυτών των διαδικασιών θεωρούμε ότι πρέπει να γίνει το συντομότερο δυνατό προκειμένου να εξασφαλιστεί η ικανότητα της Κομισιόν να δρά πολιτικά στα μέτωπα στα οποία έχουμε ανοίξει. Θεωρώ ότι με βάση το καταστατικό, το ισχύον δίκαιο, τον εσωτερικό κανονισμό έχουν ακολουθεί όλοι οι κανόνες. Οι διατάξεις του κανονισμού του προσωπικού που έχουν συμφωνηθεί μεταξύ των τριών θεσμικών οργάνων έχουν τηρηθεί στο έπακρο λαμβανομένου υπόψη ότι κάθε θεσμικό όργανο έχει υποχρέωση και δικαίωμα να ε, προσλαμβάνει τους πλέον ικανούς υποψήφιους χωρίς να ε, μπορεί ε, η κάθε απόφαση να επηρεάζεται από τις απόψεις που μπορεί να έχει κάποιο άλλο θεσμικό όργανο. Θέλω να επισέλθω σε ένα συγκεκριμένο ερώτημα. Για παράδειγμα, τι σημαίνει η μεταφορά και τι σημαίνει προκήρυξη μιας διαδικασίας μετά τη δημοσίευσή της. Τι συμβαίνει. Με βάση τον κανονισμό του προσωπικού που και εσείς έχετε ε, συμφωνήσει σε αυτόν, η Κομισιόν μπορεί όπως και τα άλλα θεσμικά όργανα είτε με μετάταξη να καλύπτει ελεύθερες θέσεις είτε μπορεί με εσωτερικές και εξωτερικές προκηρύξεις να ακολουθήσει μια άλλη διαδικασία. Και μπορώ να σας ενημερώσω ότι στα 3,5 χρόνια της θητείας της τρέχουσας Κομισιόν το Σώμα των Επιτρόπων έχει αποφασίσει σε 32 περιπτώσεις στη βάση του άρθρου 7 του κανονισμού να ε, προχωρήσουμε σε μετάταξη γενικών διευθυντών, αναπληρωτών γενικών διευθυντών, σε άλλες θέσεις. Στο ίδιο επίπεδο. Άλλοι 13 υπάλληλοι, AD 15 και 16, ε, διορίστηκαν ως ειδικοί σύμβουλοι. Και μπορώ να σας πω ότι στην ε, Κομισιόν Μπαρόζο 2 60 υπάλληλοι αυτού του βαθμού στη βάση του άρθρου 7 του κανονισμού μετατάχθηκαν. Άρα δεν έχει γίνει τίποτα το ασυνήθιστο. Ούτε για τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα, ούτε και για τα εθνικά ε, θεσμικά όργανα, υπουργεία, διοικήσεις. Κάθε φορά που έχουμε μια ελεύθερη θέση που πρέπει να καλυφθεί, αποφασίζουμε ως σώμα των επιτρόπων, ε, επιτρόπων έπειτα από εισήγηση του, του αρμόδιου επιτρόπου, αν θα προχωρήσουμε σε προκήρυξη ή σε μετάταξη για την κάλυψη αυτής της ελεύθερης θέσης. Με αυτόν τον τρόπο μπορούμε στη βάση των καθηκόντων αλλά και λαμβανωμένου υπόψη ε, του χρονικού περιορισμού και της χρονικής πίεσης ποια είναι η ορθότερη απόφαση ποιος είναι ο καταλληλότερος για την κάθε θέση. Και μπορώ να σας πω από την εμπειρία μου στα πέντε χρόνια που είχα υπό την ευθύνη μου το και της ενέργειας ότι... Ε, έλαβα έναν διευθυντή μέσω μετάταξης που ήρθε από την Γενική Διεύθυνση Γεωργίες στην Γενική Διεύθυνση Ενέργειας ακριβώς επειδή υπήρχε χρονική πίεση ε, για ζητήματα εσωτερικής αγοράς και υποδομών γι' αυτό και χρειαζόμασταν έναν κατάλληλο υποψήφιο τον οποίο και βρήκαμε και μετατάχθηκε και με αυτόν τον τρόπο ο Γενικός Διευθυντής μου που ήταν ε, ο Γενικός Διευθυντής που είχα υπό την ευθύνη μου ε, ε, μετατάχθηκε από το Κοινό Κέντρο Ερευνών στην Γενική Διεύθυνση Ενέργειας. Θέλω να πω ότι προσωπικά σε δύο περιπτώσεις έχω λάβει αντίστοιχες αποφάσεις οι οποίες μάλιστα δικαιώθηκαν από την πραγματικότητα. Τα τελευ... Τις εβδομάδες λοιπόν τέθηκαν ερωτήματα για το αν η Κομισιόν ή αν εγώ προσωπικά συμμετείχα και ήμουν ενήμερο. Επαναλαμβάνω, επειδή θεωρείτε κι εσείς ότι το θέμα αυτό είναι σημαντικό. Αυτό το πακέτο πολλαπλών θέσεων υψηλόβαθμων αξιωματούχων ήμουν ενήμερος και ακριβώς επειδή δεν συζητάμε κάθε εβδομάδα για αυτά τα θέματα αλλά για ε, την κάθε περίπτωση ξεχωριστά ε, προσπαθώντας να εξασφαλίσουμε καταλληλότητα των υποψηφίων και ε, γεωγραφική ισορροπία. Και κάπως έτσι, και έτσι μάλλον λαμβάνουμε τις αποφάσεις μας. Στο πλαίσιο λοιπόν αυτής της διαδικασίας που ακολουθήθηκε συμμετείχαμε και εγώ και το επιτελείο μου από την αρχή ε, συζήτησα και συνεδρίασα και με τους άλλους υποτελείους επιτρόπους, ε, έκανα συνέντευξη με όλους τους υποψήφιους και στη συνέχεια πριν από την λήψη απόφασης από την Κομισιόν, εγώ και ο κύριος Τίμερμανς ενημερωθήκαμε για την πρόθεση του ε, ε, Προέδρου να προαχθεί ο κύριος Ελμαϊερ με διπλή προαγωγή στη θέση του Γενικού Γραμματέα. Σε αυτό το συνολικό πακέτο λοιπόν, έπειτα από εισήγηση των αρμοδίων επιτρόπων, έγινε συζήτηση και λαμβανομένης υπόψης ε, λαμβανομένου υπόψη και του πακέτου και της πρότασης του Κομισιόν, με δική μου συγκατάθεση ομόφωνα αποφασίσαμε το διορισμό του Γενικού Γραμματέα. Πρόκειται λοιπόν για απόφαση του Σώματος των Επιτρόπων και κανείς στο Σώμα των Επιτρόπων δεν εξέφρασε αντίρρηση. Πιστεύω λοιπόν ότι τόσο η καταλληλότητα του υποψηφίου που έγινε Γενικός Γραμματέας, όσο και η διαδικασία που ακολουθήθηκε, σεβάστηκαν και το γράμμα και το πνεύμα των κανόνων. Γι' αυτό και θα ήθελα στο τέλος της σημερινή μας συζήτησης να επιβεβαιώσετε κι εσείς ότι δεν υπήρξε καμία παραβίαση του καταστατικού, του κανονισμού, του προσωπικού και ότι τα πάντα τηρήθηκαν στο έπακρο. Ευχαριστώ πολύ κύριε Επίτροπε. Θα ήθελα να δώσω το λόγο στην ε, Βαλερή Μοντεμπέλο, την οποία και έχω παρακαλέσει ε, να μας εξηγήσει τι ακριβώς προβλέπει αυτό το άρθρο 7 του κανονισμού προσωπικού. Παρακαλώ, έχετε το λόγο. Σας ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Σας ευχαριστώ που καλέσατε την νομική υπηρεσία και που μας δίνετε έτσι τη δυνατότητα να γνωμοδοτήσουμε με τρόπο αντικειμενικό και ανεξάρτητο. Καταρχάς θα ήθελα να σας πω ότι τα πράγματα δεν είναι τόσο απλά, γιατί έχουμε το καταστατικό αφενός, αλλά και τις αποφάσεις του δικαστηρίου, την ομολογία δηλαδή, και αυτά θα πρέπει να τα δούμε από κοινού. Αντιμετωπίσουμε μια κατάσταση μετάθεσης, μετάταξης ενός υπαλλήλου και πρέπει να δούμε εδώ πέρα ποιος παίρνει την απόφαση για τη μεταφορά, ποιος παίρνει την απόφαση για την απόσπαση, για, την, για τον νέο αυτοδιορισμό. Πρόκειται για τις διοικητικές αρχές των θεσμικών οργάνων και οι δικαστές πολλάκις έχουν πει ότι ουσιαστικά έχουν ε, μία ευρεία δυνατότητα εκτίμησης στα πλαίσια των ε, αποστολών που προβλέπονται. Αλλά θα πρέπει κάθε φορά να προέχει το συμφέρον της κάθε υπηρεσία και μια ισοτιμία, αντιστοιχεία ανάμεσα στις διαφορετικές θέσεις. Ποιος αποφασίζει και ποιος ελέγχει, ποιο, ποιος καθορίζει τελικά το συμφέρον της υπηρεσίας. Η έννοια αυτή είναι καθοριστική όμως, γιατί βάσει της έννοιας αυτής μπορούμε να μεταθέσουμε έναν υπάλληλο χωρίς να προκηρύξουμε τη θέση αυτή. Το συμφέρον λοιπόν τη υπηρεσία το ελέγχουν οι δικαστέ του δικαστηρίου. Αν γίνει προσφυγή βέβαια προ αυτού. Και στην περίπτωση αυτή εξετάζονται τα πραγματικά περιστατικά, τι έχει όντω συμβεί, αλλά και τι περιστάσει. Προκειμένου να σε θέση πραγματικά να εκτιμήσουν αν όντω τα όσα έχουν συμβεί συμμορφώνονται με τον κανονισμό υπηρεσιακή κατάσταση των υπαλλήλων τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Τι είναι η μετάθεση, τι είναι η μετάταξη. Η μετάθεση είναι μία μεταφορά, mutation στα γαλλικά, η μεταφορά ουσιαστικά ενό υπαλλήλου από μία θέση σε μία άλλη θέση. Ήδη από το 1981 στην απόφαση Κίντερμαν κατά Ευρωπαϊκής Επιτροπής ορίστηκε όρος αυτός, μετάθεση, και βέβαια πάντα μετάθεση έχει να κάνει με μία θέση που έχει χειρεύσει. Το ίδιο, ο ίδιος ο κανονισμός πρεσιακής κατάστασης το λέει αυτό και είναι πάρα πολύ σημαντική και η έννοια της καινής αυτής θέσης. Και αυτό διότι ορισμός, ο διορισμός ενός υπαλλήλου έχει ως μοναδικό στόχο και το λέει αυτό το καταστατικό να ανταλάβει μία καινή θέση. Αυτό είναι ο στόχος. Θα μπορούσατε να διαβάσετε το άρθρο 7 σε συνδυασμό με το άρθρο 4 του Κανονισμού Υπηρεσιακής Κατάστασης των Υπαλλήλων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι κενές λοιπόν αυτές θέσεις θα πρέπει να προκυρήσονται ή δύναται να μην προκυρήσονται. Εκεί έγκυται πραγματικά το ερώτημα. Η απάντηση είναι καταφατική. Επί της αρχής δηλαδή, το θεσμικό όργανο αποφασίζει να καλύψει την κεντή αυτή θέση και αυτή τη στιγμή παίρνει μια τέτοια απόφαση γιατί θα μπορούσε να καταργήσει και τη θέση αυτή. Αυτή τη στιγμή αποφασίζει όμω να καλύψει τη θέση, θα πρέπει να τη δημοσιεύσει. Το λέει αυτό το άρθρο 4 του κανονισμού υπηρεσιακή κατάσταση. Κάθε θέση η οποία χειρεύει και η οποία πρέπει να καλυφθεί αποτελεί αντικείμενο δημοσίευση, προκήρυξη. Υφίστανται παρεκκλήσεις ή εξαιρέσεις στη βασική αυτή αρχή. Αυτό είναι ένα ακόμα σημαντικό ερώτημα. Ναι, υπάρχουν και αυτό πρέπει να το πούμε. Εδώ πέρα θα πρέπει πραγματικά να σας δώσουμε μια αντικειμενική αξιολόγηση των πραγμάτων. Υφίστανται οι παρεκκλήσει αυτέ, αλλά δεν συμπεριλαμβάνονται στον κανονισμό υπηρεσιακή κατάσταση. Είναι παρεκκλήσει οι οποίε προκύπτουν από την ομολογία του Δικαστηρίου τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Εμεί σε 75 διαφορετικές περιπτώσεις μεταθέσεων είδαμε ότι ήταν όντως δυνατό να μεταφερθεί, να μεταταχθεί ένας υπάλληλος χωρίς να έχει προκηρυχθεί η θέση στην οποία πηγαίνει, χωρίς να δημοσιευθεί δηλαδή η θέση αυτή, στην ε, περίπτωση της ε, επανακάλυψης της θέσης αυτής, της ε, απόσπασης του υπαλλήλου αυτού προς μία άλλη θέση. Να δώσω περισσότερες εξηγήσεις ο υπάλληλο ε, σε κάθε περίπτωση μεταφέρεται στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων του. Σας παραπέμπω σε μια απόφαση που είναι σημαντική, Ράσμουσεν κατά Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Ουσιαστικά ο υπάλληλος ε, μετακινείται με την εργασία του, με τις αρμοδιότητες τις οποίες έχει. Επίσης, στα πλαίσια της παρέκκλησης αυτής, η οποία θα πρέπει να εφαρμόσετε βέβαια με τρόπο ιδιαίτερα περιορισμένο, οι δικαστές είπαν ότι μια τέτοια μετάθεση, μεταφορά θα πρέπει να αιτιολογείται από το ίδιο το συμφέρον της εν λόγω οικίας υπηρεσίας. Τι σημαίνει αυτό στην πράξη. Ότι η κατάσταση πρέπει να είναι αρκετά σοβαρή, αρκετά επίγουσα και ότι αυτό θα πρέπει να επιβεβαιώνεται στις περισσότερες περιπτώσεις. Σα είπα ότι προκειμένου να προτιμάσω τη σημερινή μου παρέμβαση εξέτασα την νομολογία του Δικαστηρίου τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Εργάστηκα πολύ λοιπόν αυτό το Σαββατοκύριακο. Εξέτασα 75 διαφορετικέ υποθέσει που εκδίκασε το δικαστήριο όσον αφορά τέτοιε περιπτώσει μεταθέσεων. Έχουμε τρία διαφορετικά είδη καταστάσεων που μπορούν να προκύψουν επί των οποίων έχουν αποφανθεί δικαστές. Έχουμε την περίπτωση του υπαλλήλου που μετακινείται με το πόσο του, με εργασία του ουσιαστικά, όταν ε, βρίσκεται σε μια ιδιαίτερα ε, δύσκολη κατάσταση, σε μια τεταμένη κατάσταση εργασίας. Στην περίπτωση Μπεν ε, κατά Ευρωπαϊκό Κοινοβουλίο έχουμε μετάταξη ενός υπαλλήλου, ο οποίος ήταν θύμα παρενόχλησης. Αυτή ήταν η πρώτη περίπτωση. Μία άλλη περίπτωση που έχει προκύψει και που την έχουμε σε πολλέ υποθέσει που έχει εκδικάσει στο δικαστήριο είναι ένα υπάλληλο ο οποίο μεταφέρεται, μετατίθεται όταν υπάρχουν κάποιε αμφιβολίε όσον αφορά κάποιε παρατυπίε και ότι είναι πολύ δύσκολο τελικά να αποφασίσει κανεί αν θα πρέπει να κάνει μία έρευνα ή όχι. Αναφέρομαι εδώ πέρα στην υπόθεση κλωτου κατά Ευρωπαϊκή Επιτροπή, υπόθεση που έχει εκδικάσει το Δικαστήριο τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Και τέλο και πιο σημαντικό θεωρώ ο υπάλληλο μπορεί να μετατεθεί όταν είναι αναγκαίο να οργανωθεί ή να επαναργανωθεί η υπηρεσία, ακριβώς επειδή κρίνεται ότι η υπηρεσια ακριβω επειδη κρινεται αυτή δεν λειτουργεί με το βέλτιστο δυνατό τρόπο. Στην περίπτωση αυτή, ο δικαστή εξετάζει την υπόθεση με πολύ μεγάλη σύνδεση και προσοχή, θα λάβει υπόψη του τα καθήκοντα της υπηρεσίας, τις αρμοδιότητες προβλέπονται στα πλαίσια τη υπηρεσία, καθώ επίση και την ε, ιεραρχική ε, δομή μια σχετική απόφαση που έχουμε εδώ πέρα είναι η απόφαση στην υπόθεση Guggenheim κατά Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Στην απόφαση αυτή έχουμε το Ευρωπαϊκό Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης, το οποίο εδράζεται στην ε, Θεσσαλονίκη και όπου ο δικαστής είχε αποφασίσει ότι όντω από νομικής πλευράς θα μπορούσαν να μετατεθούν πολλοί υπάλληλοι σε σημαντικές οργανικές θέσεις χωρίς να προκηρυχθούν οι θέσεις αυτές και αυτό προκειμένου να επαναδιοργανωθεί η όλη υπηρεσία. Αλλά βέβαια λέει δικαστής ότι η συνήθις διαδικασία και η πιο κατάλληλη διαδικασία τελικά θα ήταν να είχαν προκηρυχθεί και δημοσιευθεί οι θέσεις αυτές. Το βασικό κριτήριο λοιπόν του δικαστή είναι να έχουμε κάθε φορά ικανούς υπαλλήλους του πλέον αρμόδιου υπαλλήλου, Αυτό άλλωστε το λέει και ο κανονισμό υπηρεσιακής κατάστασης. Και για αυτόν τον λόγο θα πρέπει να προβλέπετε μια εσωτερική διαδικασία επιλογή, Αυτό είναι δικαστή στην υπόθεση Guggenheim. Μπορούμε να οργανώσουμε μια εσωτερική διαδικασία επιλογή χωρί να έχουν προκηρυχθεί κάποιε θέσει. Ο δικαστή μα λέει πω ναι, είναι δυνατό, μπορούμε σε εσωτερικό επίπεδο να κάνουμε συγκριτική αξιολόγηση των ε, αρμοδιοτήτων, των προσόντων μάλλον, των υποψηφίων και εν συνεχεία μπορεί να αποφανθεί κανείς για το ποιος είναι ο πλέον κατάλληλος. Συνοψίζοντας λοιπόν η αρχή του άρθρου 7, όπου προβλέπεται ότι θα πρέπει να γίνεται δημοσίευση της θέσης, συνοδεύεται από τις δυνατότητες παρέκκλησης που προβλέπει το δικαστήριο, αρκεί η μετάταξη, η μετάθεση του υπαλλήλου, η οποία μπορεί να γίνει χωρίς προκήρυξη, αιτιολογείται δεόντως για λόγους συμφέροντος της ίδιας υπηρεσίας. Ευχαριστώ πολύ για τις πληροφορίες αυτές. Συμπέρασμα λοιπόν που κρατάω εγώ είναι να, ότι θα ήταν καλύτερο να είχε υπάρξει προκήρυξη και Βεβαίω το γεγονό ότι κάτι τέτοιο δεν συνέβη προκύπτει και από τι απαντήσει που δόθηκαν στι ερωτήσει μα. Λοιπόν, θα ήθελα τώρα, όπω συμφωνήσαμε, να δώσω πέντε λεπτά σε, στους συντονιστές των πολιτικών ομάδων. Ε, θα κάνουμε τη διαδικασία του Pink pong Πέντε λεπτά δηλαδή για ερώτημα και απάντηση. Ο κύριος Σάβαμα έχει το λόγο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Πολλά έχουν ε, συζητηθεί στους διαδρόμους Ευρωπαϊκή Ένωσης αλλά και στα ΜΜΕ και έχει προκληθεί αρκετός εκνευρισμός και ανησυχία. Οπότε είναι ξεκάθαρο ότι θα πρέπει εμεί να διασκεδάσουμε αυτές τις ε, εντυπώσεις και αμφιβολίες και γι' αυτό ευχαριστούμε κύριε Επίτροπε που ήρθατε στην Επιτροπή μας για να μας βοηθήσετε να ξεκαθαρίσουμε το τοπίο. Θέλω τώρα να σας πω το εξή για να είμαστε σαφείς. Χρειαζόμαστε 100% διαφάνεια και θα πρέπει επίσης να προσέξουμε ιδιαίτερα στο θέμα της ακυριότητος ε, στα πιο υψηλά επίπεδα των θεσμικών οργάνων. Άρα το ερώτημα που αναδύεται είναι κατά πόσον η έλλειψη της διαφάνειας σε αυτή την περίπτωση, δηλαδή όσον αφορά την δικασία του διορισμού του κ. Σελμάγερ, εάν έγινε ελλείψη ή τέλο πάντων σε παραβίαση αυτή τη υποχρέωση τήρηση της ηθική ακυριότητα και τη ε, διαφανείας. Δυστυχώς οι ενδείξεις εκεί μα οδηγούν. Επίση υπάρχει και κάτι άλλο που αντιβαίνει στην ε, ηθική ακυριότητα. Υπάρχει κάποια επικάλυψη δηλαδή, των δύο αρχών, δηλαδή ε, το, το ένα πράγμα οδήγησε στο άλλο. Ακριβώ αυτό και διερευνούμε. Αυτό είναι και το καθήκον μας. Οπότε έχω δύο ερωτήσει, ε, κύριε Έτιγκερ. Η πρώτη είναι η εξή. Τηρήσατε όλους τους προβλεπόμενους κανόνες κατά τη διαδικασία, ούτως ώστε να μην υπάρχει καμία σκιά για το νόμιμο του διορισμού. Και το δεύτερο, πολύ σημαντικό για μένα, εσείς ως ο αρμόδιος για το προσωπικό επίτροπος, πώς Αξιολογείται αυτήν την διαδικασία. Νομίζω ότι κύλησε εύρεθμα όπως θα έπρεπε να εξελιχθεί. Κύριε Επίτροπε, παρακαλώ. Κύριε Προβουλευτά, κυρίε και κύριοι, Ελέγχοντας όλα τα βήματα που ακολουθήθηκαν, καταλήξαμε στο συμπέρασμα ότι τηρήθηκαν όλοι οι ισχύοντες κανόνες. Και ότι οι διατάξεις στις οποίες εσείς έχετε καταλήξει και εσείς έχετε θεσπίσει χαρακτήρισαν τη διαδικασία αυτή. Το αν η διαδικασία αυτή ήταν εύρυθμη ή λειτουργήσε καλά, δεν είναι, δεν είναι νομικό το ερώτημα αυτό, είναι πολιτικό ή και προσωπικό το ερώτημα. Θα μπορούσαμε βεβαίω όλοι να εξετάσουμε τι θα μπορούσαμε να είχαμε κάνει και καλύτερα. Γιατί φυσικά εκ των υστέρων όλοι μας είμαστε σοφότεροι. Ξεκινώ από την Κομισιόν και σας λέω ότι αφού σας αποστήλαμε την Κυριακή το πρωί τις απαντήσει μα. έγκυται σε εσάς να αξιολογήσετε τη διαδικασία και το αποτέλεσμα αυτής. Γι' αυτό και είναι απαραίτητο ένα χθεσινό tweet εκπροσώπου να αποσυρθεί. Ακριβώς γιατί δεν αντεποκρινόταν στην καλύτερη, στην, ε, στην, ε, στις απόψεις της Κομισιόν. Το ερώτημα λοιπόν ε, δεν απευθύνεται στην Κομισιόν στην πραγματικότητα, απευθύνεται σε εσά τους ίδιους. Εσείς λοιπόν έχετε ευθύνη να μας πείτε αν θεωρείτε, αν, πώς και πού παραβιάστηκαν κανόνες. Και από εκεί και πέρα να γίνει αυτή η συζήτηση. Και ταυτόχρονα θέλω να δηλώσω το εξής. Φυσικά, στην πολιτική και στη δημόσια σφαίρα πρέπει κανείς να είναι έτοιμος να δεχτεί και επιθέσεις. Αυτό αφορά εσάς, αφορά εμένα προσωπικά, αφορά όλους μας. Όμως η μεταχείριση την οποία, ε, η οποία επιφλάχθηκε στο Μάρτιν Σέλμαϊρ, για την οποία μπορεί κανείς να έχει τη μία ή την άλλη άποψη. Και οι πολύ άσχημες επιθέσεις που δέχτηκε δεν θεωρώ ότι είναι χρήσιμες. Κάτι τέτοιο δεν περιποιεί τιμή ούτε στο Κοινοβούλιο, ούτε στην Κομισιόν. Θα μπορούσα να σας δώσω και ένα-δυο άλλα παραδείγματα, όπου θα μπορούσα ενδεχομένως εκ των υστέρων γνωρίζοντας τα πράγματα να είχα λάβει μια διαφορετική απόφαση. Όμως, με βάση ε, τα όσα γνωρίζουμε και τα όσα έχουμε ελέγξει διεξοδικά, δεν ε, ούτε ένας κανόνας. Η κυρία Γιάλα Σέντερ έχει το λόγο. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε αλλά και τον Επίτροπο που δέχθηκε να έρθει εδώ για αυτή την ακρόαση. Απλώς θα ήθελα να σας πω ότι όπως είπατε και εσείς για την εφαρμογή των κανονών έχουμε πάντοτε το γράμμα και το πνεύμα. Και εδώ για τόσες βδομάδες εξετάζουμε εδώ το καλό και το κακό, τις συνθήκες που περιβάλλουν αυτή την πράξη και τελικά βλέπουμε ότι όσα γίνανε δεν ανταποκρίνονται στο πνεύμα του νόμου. Τρία έχω να αναφέρω προς εσάς Πρώτα πρώτα ο επικεφαλής του ιδιαίτερου γραφείου. Από ό,τι φαίνεται ήταν η μας ευθύς εξ αρχής. Και λέγεται ότι επίσης ενημερώθηκε τη στιγμή που έγινε η αλλαγή. Όμως προκύπτει ότι υπήρξε ενημέρωση και αρχές του 2018 αλλά δεν προκύπτει αν υπήρχε ενημέρωση πριν τις 20 Φεβρουαρίου για τον κύριο Ταλιάνερο ο οποίος είχε ενημερωθεί και ότι πρόκειτο να αποχωρήσει από αυτή τη θέση Οπότε έχουμε εδώ πέρα μία σκιά σύγκρουση συμφερόντων, αλλά επίσης και παραβίαση του καθήκοντος εμπιστοσύνη για τις πληροφορίες που δόθηκαν. Οπότε βλέπουμε ότι ήταν στο βιβλιογραφείο αυτός ο κύριος και δεν ξέρουμε κατά πόσον τηρήθηκαν όσα έπρεπε όσον αφορά λοιπόν την διαφάνεια. Και αυτή η υποψήφια αποθαρρύνθηκε όταν ήρθε η ώρα της αξιολόγησής της από τους αξιολογητές την απεθάρρυναν. Πώς ακριβώς παρετήθηκε. Με επιστολή. Επίσης έχουμε αυτό το, το, φάκελο με τους διορισμούς και είχαν αντίθεση, είχαν ένσταση, αισθάνθηκαν ταπεινωμένοι οι γενικοί διευθυντές και μας είπατε το αναλάβατε εσείς κύριε Επίτροπε μήπως θα πρέπει κάπως να αλλάξουν οι κανόνες και να υπάρχουν διαφορετικές συνθήκες, να υπάρχει ισότητα ευκαιριών, να υπάρχει πραγματικά συλλογική προσπάθεια και συλλογική διαδικασία που να οδηγεί στον ε, διορισμό ούτω ώστε να τηρείται όχι μόνο το γράμμα αλλά και το πνεύμα του νόμου. Επίσης, σύμφωνα με το άρθρο 20, συμφωνείται στο τέλος της εντολής ε, στο τέλο της εντολή τη θητεία τη Επιτροπή Γιούνκερ να αναφέρουμε τα σχετικά με το Γενικό Γραμματέα. Επίτροπε. Äh, δεν, κατάλαβα ε, μία από τις παρατηρήσεις σας. Είπατε κάτι για κομματικές ε, ε, συνεδριάσεις, ίσως δεν κατάλαβα. Εγώ δεν έχω υπόψη μου καμία κομματική συνεδρίαση όπου ε, ο φάκελος των ε, υποψηφίων να συζητήθηκε, πόσο μάλλον η θέση του Γενικού Γραμματέα ή να τέθηκε υποδιαπραγμάτευση ε, ο διορισμός ε, και η υποψηφιότητα αυτή. Δεύτερον, δεύτερη υποψήφια για την προκηρυχθήσα θέση του αναπληρωτή Γενικού Γραμματέα υπήρξε πράγματι, πήγε στο Assessment Center, στο κέντρο αξιολόγησης, θεωρήθηκε Όμω, όχι ότι δεν έχει τι ικανότητε, μόνη τη απέσυρε την υποψηφιότητά τη. Είχε ξεκινήσει την υποψηφιότητά τη, πράγματι, είχε υποβάλει αίτηση, αλλά στη συνέχεια την απέσυρε. Δεύτερον, αν πρέπει να αλλάξει κάτι στη διαδικασία διορισμού Γενικού Γραμματέα. Βεβαίω, το να κάνουμε συζητήσει για βελτίωση των διαδικασιών προσλήψεων, φυσικά αυτό είναι κάτι που είναι πάντοτε ένα θέμα ανοιχτό. Και αυτό αφορά την Κομισιόν, το Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο όλα τα θεσμικά όργανα της Ένωσης. Και είπατε, κυρία Σέντερ, ότι τηρήθηκε μεν το γράμμα των κανόνων. Εγώ αυτό θεωρώ ότι είναι ήδη κάτι ικανοποιητικό. Άρα δεν συζητούμε αυτό. Διότι σε τελική ανάλυση οι κανόνες και οι νόμοι που καταρτίζει και θεσπίζει το Κοινοβούλιο αποτελούνται από κείμενα. Από λέξεις, από παραγράφους, προτάσεις και γράμματα. Αυτά διαβάζουμε, αυτά ερμηνεύουμε, αυτά τηρούμε. Αν λοιπόν έχει τηρηθεί το γράμμα του νόμου, αυτό ήδη διασκεδάζει ανησυχίες και αμφιβολίες που έχουν εκφραστεί σε σχέση με τη διαδικασία που ακολουθήθηκε. Είπατε όμως ότι το πνεύμα των κανόνων ενδεχομένως δεν τηρήθηκε, στο έπακρο τουλάχιστον. Αν λοιπόν θεωρείτε ότι έστω εν μέρη ε, τηρήθηκε το πνεύμα, έχετε πει ότι τηρήθηκε 100% το γράμμα και εν μέρη το πνεύμα του κανόν, των κανόνων. Θα ήθελα όμως να μου εξηγήσετε τι ακριβώς εννοείτε. Υπάρχει κάποια απόκληση μεταξύ του γράμματος και του πνεύματος του νόμου. Γιατί αν θεωρείτε κάτι τέτοιο, αν πιστεύετε κάτι τέτοιο, τότε πρέπει ενδεχομένως να αλλάξουμε το γράμμα. Εγώ, όπως είπα, είμαι νομικός. Διότι το να μου λέτε ότι κατά την δική σας ερμηνεία δεν τηρήθηκε το πνεύμα του κανόνα, τότε αυτό δεν με βοηθάει ιδιαίτερα. Διότι υπάρχει κανονισμός προσωπικού, ο οποίος διέπει τις προσλήψεις και τους υπαλλήλους την εργασία των υπαλλήλων τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Αν θεωρείτε ότι αυτά πρέπει να αλλάξουν, αν, αν θεωρείτε ότι πρέπει ο κανονισμό αυτό να αλλάξει, παρακαλώ, είμαστε στη διάθεσή σας. Αυτό εσεί το είπατε. Εγώ να το δεχτώ, εάν μου απαντήσετε για το τι έγινε ακριβώ τότε που λέει early 2018, το 2018 στην αρχή δηλαδή, που είπε η κυρία Ταλιάνερ ότι πρόκειται να εγκαταλείψει την Γενική Γραμματεία. Και αν μίλησε ο κ. Γιούνκερ με τον επικεφαλής του ιδιαίτερου του γραφείου τότε. Εγώ πιστεύω ότι έτσι έγινε και γι' αυτό είχαμε αυτή την ε, ε σύγκρουση ε, ε, συμφερόντων και επίσης ε, την παραβίαση του απορρίτου των πληροφοριών εκείνων. Οπότε αυτό πρέπει να μα Εάν η κυρία τα μέρωσε ενημέρωσε αρχές του 18 τον κύριο Γιούγκερ <clears throat> και ακριβώς πότε αυτό το early 2018 τι πάει να πει. Και επίσης αυτές οι πληροφορίες διαβιβάστηκαν πριν στις 20 του μηνός οπότε είχαμε τα επίμαχα γεγονότα γιατί αυτό μας είπε η τέλος πάντων αυτά αρνήθηκε σε σχέση με τις ε, ληφθείς αποφάσεις. Αν όλα αυτά να γίνανε τυχαία, από σύμπτωση. Δεν θέλει το Κοινοβουλίο να ψεύδεται η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Άρα πρέπει να μάθουμε ακριβώς με ποιο τρόπο ο επικεφαλής του ιδιαίτερου Γραφείου, ο οποίος αναγνωρίζει ότι ε, δέχθη αυτές τις ε, πληροφορίες. Εάν επομένως ε, έλαβε γνώση πριν ληφθούν οι σχετικές αποφάσεις. Επίτροπο κύριοι βουλευτέ, από πολυέρθμε συζητήσει που είχα και από την εξέταση των εγγράφων, μπορώ να σας πω ότι έχω σχηματίσει την εξή εικόνα. Ο επικεφαλής υποψήφιος κύριος Γιούγκερ ήταν ο μελλοντικός πρόεδρος της Κομισιόν. Όπως και στο παρελθόν είχε και ένα επιτελείο το οποίο τον προετοίμασε για την ανάλυση των καθηκόντων Όλα αυτά έγιναν τον Ιούνιο-Ιούλιο του 2014 προκειμένου να προετοιμάσει τη νέα Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Τη δομή τη στη συνέχεια έλαβε και συναντήθηκε με τους υποψηφίους των κρατών μελών. Στη συνέχεια κάποιοι από τους υποψηφίους αυτούς ελέγχθηκαν ε, με βάση ε, την καταλληλότητά του για το κάθε ε, χαρτοφυλάκιο. Χρειάστηκε βεβαίως να πει ε, σε, κάποιους, σε κάποια κρατημέλη να πει ότι ε, πρέπει να μας στείλετε γυναίκα γιατί το Κοινοβούλιο θέτει ως όρο να υπάρχουν τουλάχιστον εννέα γυναίκες επίτροποι. Επικεφαλής λοιπόν αυτής της ομάδας προετοιμασίας του κυρίου Γιούνκερ ήταν ο Μάρτιν Σέλμαϊρ. Ήταν λοιπόν από την πρώτη μέρα εκεί μαζί του και η Κάθριν Ντέι ήταν έως τότε γενικός, γενική γραμματέας, η οποία όμως είχε δηλώσει την πρόθεσή της να παρετηθεί. Γι' αυτό, για λόγους συνέχειας, χρειάστηκε να ακολουθεί η διαδικασία που ακολουθήθηκε. Εγώ, την άνοιξη του 2015, έλαβα έναν αντίστοιχο φάκελο προετοιμασίας, για την ε, αξιολόγηση και τη λήψη αποφάσεων. Και στο πλαίσιο αυτής της διαδικασίας η Κάθριν Ντέι είπε ότι θέλει να αξιοποιήσει αυτήν την διαδικασία που μια ακολουθείται προκειμένου να παραιτηθεί από τη θέση της Γενικής Γραμματέας. Η παρέτηση αυτή έγινε δεκτή από τον κύριο Γιούγκερ και στη συνέχεια με το στενότερο συνεργάτη του, το διευθυντή του γραφείου του, συζήτησε το ζήτημα της διαδοχής της. Ο Ζαν Κλοντ λοιπόν κατέληξε στο συμπέρασμα ότι θα έπρεπε με μετάταξη από, να, μεταφέρει τον, τον, ε, τον κύριο Ιταλιάνερ από Γενικό Διευθυντή και να τον διορίσει ως Γενικό Γραμματέα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Ο κύριος Ιταλιάνερ στην αρχή λοιπόν της θητείας του είχε δηλώσει ότι δεν θέλει να εξαντλήσει την θητεία του. Ότι για προσωπικούς λόγους θα παρετούνταν από τη θέση αυτή πριν από τη λήξη της θητείας της Κομισιόν και έτσι συμφωνήσαμε σε δύο ή κάτι παραπάνω χρόνια για δική του θητεία. Στο διάστημα αυτό λοιπόν ο πρόεδρος μου του ζήτησε επανειλημμένος να παραμείνει για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα ή δυνατόν έως το τέλος της θητείας της Κομισιόν, το φθινόπωρο του 19. Για παράδειγμα, στην καλύτερη περίπτωση. Και τέτοιου είδους προσπάθειες έκανε ο κύριος Γιούγκερ επανειλημμένος έως και τον Ιανουάριο του 2018. Αυτό μπορεί να σας το επιβεβαιώσει και ο κύριος Ιταλιάνερ και ο κύριος Γιούγκερ. Κάποια στιγμή όμως ήταν σαφές ότι στο Σώμα των Επιτρόπων θα συζητηθεί ο φάκελος των υποψηφιωτήτων και εκεί υπήρξε και το ερώτημα για το αν ο κύριος Ιταλιάνερ θα μείνει ή θα αποχωρήσει και ο κύριος Ιταλιάνερ αποφάσισε να αποχωρήσει. Έτσι λοιπόν ο κύριος Γιούγκερ κλήθηκε να αποφασίσει ποιος θα ήταν ο κατηλότερος υποψήφιος για τη θέση του Γενικού Γραμματέα και κατέληξε στο συμπέρασμα ότι ο κύριος Σέλμαερ είναι ο καταλληλότερος. Είναι προτίμησή του αλλά αιτιολογημένα με επιχειρήματα ως προς τα προσόντα του και την προσωπικότητά του θεώρησε ο κύριος Γιούγκερ ότι ο κύριος Σέλμαερ θα ήταν ο καταλληλότερος την ημέρα πριν από την εξέτηση, εξέταση αυτού του φακέλου υποψηφιότητων ενημέρωσε ο κύριος ε, ότι το Σώμα των Επιτρόπων, ότι ο κύριος Ιταλιάνερ θέλει να αποχωρήσει και ότι ο κύριος Γιούγκερ θέλει να προτείνει τον κύριο Σέλμαερ. Ενημέρωσε λοιπόν πρώτα τον κύριο Τίμερμανς ως πρώτο αντιπρόεδρο και ως εξαιρετικό σύμβουλο θα προσθέσω εδώ, παρά το γεγονός ότι ανήκει σε, άλλο, ε, σε άλλη πολιτική ομάδα. Τον ενημέρωσε λοιπόν ο κύριος Γιούγκερ και το βράδυ της 20ης Ιανουαρίου, όταν εγώ ε, του παρουσίασα το φάκελο των υποψηφιωτήτων που είχε προετοιμαστεί για εμένα, όταν λοιπόν του παρουσίασα τις αξιολογήσεις μου για μια σειρά από ε, προκηρύξεις, από μετατάξεις, μεταθέσεις, με ενημέρωσε σχετικά με την πρόθεσή του, δεδομένου της, δεδομένης της απαχώρησης του κύριου Ιταλιάνερ να διορίσει τον κύριο Σελμαέρ στη θέση του Γενικού Γραμματέα. Περισσότερα από αυτά δεν μπορώ να σας πω, δεν μπορώ να σας δώσω περισσότερες πληροφορίες. Από τις τελευταίες λοιπόν ευρωεκλογέ έως και σήμερα θεωρώ ότι έχουν τηρηθεί σε όλες τις περιπτώσεις οι κανόνες που ισχύουν. Thank you to the σας ευχαριστώ κύριε Επίτροπε για την παρουσία σας εδώ σήμερα. Είναι, θα έλεγα, πολύ ενδιαφέρον το ότι μιλάμε για το πώς βλέπει η κοινή γνώμη το ζήτημα. Ο Επίτροπος αναφέρθηκε σε αυτό ξαφνικά μας λέτε ότι στέλνετε τις απαντήσεις στα μέσα της νύχτας και ότι ο εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής έστειλε ένα tweet λέγοντας ότι θα πρέπει να ασχοληθούμε πλέον με πιο σοβαρά ζητήματα που δεν υπάρχει καμία παρατυπία. Μήπως περιμένετε να ζητήσουμε και συγγνώμη από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή που χάνουμε πάρα πολύ χρόνο με το ζήτημα αυτό. Υπάρχει πάντω, θα έλεγα, μια γενικότερη τάση στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή να δείχνεται μια κάποια υπεροψία για το ζήτημα αυτό από πλευρά CCR είμαστε δυσαρεστημένοι που ακόμα και σήμερα και συζήτηση που έγινε στην Ολομέλεια ο κύριος ε, Γιούνκερ δεν ε, μας ε, επεξήγησε ακριβώς ποιες είναι οι τις διαδικασίες. Καταλαβαίνω ότι τα καθήκοντά σας αυτά δεν είναι ιδιαίτερα εύκολα. Θα ήθελα παρόλα αυτά να σας θέσω και κάποια άλλα ερωτήματα αφότι ε, δεν καταφέρνουμε τελικά μέσω των προηγούμενων ερωτήσεων να φτάσουμε πραγματικά στην ουσία του πνεύματος του νόμου. Η πρώτη μου λοιπόν ερώτηση είναι η ακόλουθη. Ο κύριος ε, Σελμάιερ, πώς πιστεύετε ότι ε, προβάλλει τελικά την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ποια είναι η αντίληψη που έχει το κοινό για αυτόν, ο πλέον υψηλόβαθμο δημόσιος υπάλληλος στα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα πηγαίνει σε πολιτικά κόμματα του δικού σας του κόμματος και του κόμματος του κυρίου Γιούνκερ. Θεωρείτε ότι είναι θεμητός τρόμος αυτός προκειμένου η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να ανακτήσει την εμπιστοσύνη των Ευρωπαίων πολιτών στην Ευρωπαϊκή Δημόσια Διοίκηση. Δεύτερο ερώτημα. Θεωρείτε ότι ακούσαμε μάλλον ότι ο κύριος Γιούνκερ είπε ότι θα παραιτηθεί και αυτός αν χρειαστεί να παραιτηθεί ο κύριος Σέλμαϊερ πραγματικά αξιοσημείωτη δήλωση αυτή, αν όντω αληθεύει. Στην πράξη, τι σημαίνει η δήλωση αυτή του κύριου Γιούνκερ, συμπεριλαμβάνει και την παρέτηση άλλων επιτρόπων του συντόλου τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Πώ θα πρέπει να αξιολογήσουμε όλη αυτή τη ρητορική από τον πρόεδρο τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ο Επίτροπο. Επιτρέψτε μου, κύριε Ευρωβουλευτά, να σας απαντήσω ξεκάθαρα. Πρώτον, βρίσκομαι εδώ ακριβώς γιατί θεωρώ ότι το θέμα αυτό είναι σημαντικό και σοβαρό. Γνωρίζω τις διαδικασίες που ακολουθείτε στο Κοινοβούλιο, γνωρίζω τις διαδικασίες που ακολουθούνται στην Κομισιόν και γι' αυτό μπορώ να σας ε, επιβεβαιώσω ότι ακολουθήθηκαν νόμιμα όλες τις διαδικασίες. Είμαι στη διάθεσή σας και μετά τη σημερινή μας συζήτηση, σημερινή να ε, προχωρήσω σε περαιτέρω απαντήσεις σε ερωτήματα αν έχετε. Εγώ διάβασα επίσης για αυτήν την κομματική εκδήλωση. Περί σε πρόκειτο. Όπως κάθε φορά πριν από σύνοδο κορυφής υπάρχουν συναντήσεις κομματικών ηγεσιών. Ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος, Γιώζεφ Ντόλ, συγκάλεσε λοιπόν μια τέτοια συνεδρίαση. Σε αυτήν συμμετείχε και ο Αντώνιο Ταγιάννη, που επίσης ανήκει στο ΕΛΚ και ο πρόεδρος της ε, Κομισιόν και ο κύριος Τούσκ. Όλοι αυτοί λοιπόν ακολουθούνται στο, ε, και συνοδεύονται πηγαίνοντας στο κτίριο του Συμβουλίου. Και το ερώτημα ήταν ποια θα είναι η αντίδραση που θα δοθεί στα τελωνιακά και εμπορικά μέτρα που ε, επρόκειτο να λάβουν οι Ηνωμένε Πολιτείε της Αμερικής. Ο κύριος Σέλμαϊρ λοιπόν παρακολούθησε, ε, βρισκόταν μάλλον στο κτίριο, δεν συμμετείχε όμως σε αυτήν την κομματική συνάντηση βρισκόταν έξω από την αίθουσα, όπως και άλλοι διευθυντές πολιτικών γραφείων, διευθυντές γραφείων πρωθυπουργών, αρχηγών κρατών και κυβερνήσεων. Η συνοδεία λοιπόν μένει στο διάδρομο, έξω, όμως μπορεί, εφόσον χρειαστεί, να προβεί σε διαπραγματεύσεις, σε παροχή συμβουλών, καθώς ε, η κυρία Μάλστρομ βρισκόταν στην πτήση επιστροφής της από τις ΗΠΑ προκειμένου να δοθεί η καλύτερη δυνατή απάντηση ως Ευρωπαϊκή Ένωση σε αυτές τις απειλές περί ε, θέσπισης ε, αρνητικών, εμπορικών και τελωνιακών δασμολογικών μέτρων από τις ΗΠΑ. Δεν θεωρώ λοιπόν ότι ήταν μεμπτό το γεγονός ότι ο κύριος Σέλμαϊρ βρισκόταν στο κτίριο όπου διεξεγόταν η Σύνοδος Κορυφής ακριβώς διότι ρόλος του είναι να παρέχει συμβουλές σε περιπτώσεις όπου ε, χρειάζεται. Τώρα για το ποια είναι η δημόσια εικόνα. Η εικόνα στην κοινή γνώμη. Δεν έχουμε να κάνουμε μόνο με τη φούσκα των Βρυξελών. Το θέμα αυτό αφορά τους πολίτες που ενδιαφέρονται για την πολιτική και εκτός Βρυξελών. Γι' αυτό και η σοβαρότητα του θέματος είναι τόσο υψηλή. Η δημόσια αντίληψη και η εικόνα που έχει σχηματιστεί δεν είναι θετική. Όμως, παράκληση από την πλευρά μου. Αν όλοι μας θέλαμε η εικόνα αυτή να είναι τουλάχιστον αντικειμενική, τότε νομίζω ότι όλοι μας μπορούμε να κάνουμε την αυτοκριτική μας, να αξιολογήσουμε ποια θα ήταν η καταλληλότερη και πλέον ενδεδειγμένη ε, διαδικασία που θα έπρεπε να είχε ε, ακολουθηθεί. Ο κύριος Γαμπράντη. Yeah. <clears throat> Ε, πρόεδρε, ευχαριστώ. Από όλα όσα ακούσαμε μέχρι τώρα του Επιτρόπου, μπορούμε να πούμε ότι από ό,τι φαίνεται τις τελευταίες εβδομάδες και μήνες γινόμαστε μάρτυρες ενός θεατρικού έργου με τη βάση ενός σεναρίου από τον πρώτο της Επιτροπής, από τον κ. Σέλμαν, αλλά κανείς δεν το έχει διαβάσει αυτό το σενάριο και έχουν ρόλους και 27 υπόλοιποι επίτροποι. Ε, αυτό δεν έχει καμία σχέση με το ότι έχει να κάνει με την ε, ακυριότητα. Και είπαμε όμως ότι τελικά το κοινοβούλιο και οι δημοσιογράφοι δεν έπαιξαν το ρόλο του σύμφωνα με το σενάριο. Αυτό είναι κάτι σαν πραξικόπημα πολιτικό και διοικητικό. Και έχω να ρωτήσω τον κύριο Τιγκέρ το εξή. Αντιλαμβάνομαι ότι ο πρόεδρος Γιούνκερ είμαι βέβαιος μάλλον ότι είπε στον κύριο Σελμάρ για την αποχώρηση του κύριου Ταλιάνη, αλλά δεν καταλαβαίνω γιατί δεν το είπε και στον κύριο Έτιγκερ που είναι ο αρμόδιος επίτροπος. Τι θα πει αυτό, έλλειψη εμπιστοσύνη από πλευρά Προέδρου τη Επιτροπή προ τον αρμόδιο για το προσωπικό επίτροπο. Δεν θεωρείτε ότι σας παρέκαμψε κύριε Έντιγκερ Δεν θα έπρεπε να σας τα πει ταυτόχρονα όταν τα είπε στον κύριο Σελμάκη εδώ και δύο χρόνια. Είχε εξαγγείλει ο κύριος Γιούγκερ ότι θέλει πολιτική επιτροπή με πολιτικές αποφάσεις. Να, τώρα έχουμε ένα τέτοιο παράδειγμα, πολιτικές απόφασεις με πολιτικές επιπτώσεις. Είναι πάρα πολύ σημαντικές οι επιπτώσεις. Έχει αμαυρωθεί πάρα πολύ η εικόνα και η αξιοπιστία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και τα όσα μας απαντούν στα ερωτήματά μας είναι σαν αυτά που απαντάει ο Τραμπ σε αντίστοιχε κατηγορίες. Όλα αυτά θα στιγματίσουν, θα κουκουλώσουν κατά κάποιο τρόπο τις ευρωπαϊκές εκλογές. Μα τι θα κάνει το σώμα των επιτρόπων, θα κάνει κάτι για να αποκαταστήσει τα πράγματα, κύριε Επίτροπε. Ε, ε, Η διαδικασία αντικατοπτρίζει όχι μόνο τους εσωτερικούς ε, κανόνες, αλλά και τους ευρωπαϊκούς κανόνες. Ο κανονισμός προσωπικού δηλαδή, στις δημόσιες διευλεύσεις που έγιναν και στον οποίο κατέληξαν Συμβούλιο και Κοινοβούλιο και που εφαρμόζεται έκτοτε σε όλες τις προσλήψεις στα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα. Δεύτερον, εγώ δεν θα έκανα λόγο για πραξικόπημα. Όποιο γνωρίζει τι θα πει πραξικόπημα και όποιο φιλομετρήσει και κανένα ένα ε, ιστορικό βιβλίο για τον 20ο αιώνα, για παράδειγμα, στην Ευρώπη, θα καταλάβει ότι η έννοια αυτή έχει μια τελείως ε, διαφορετική ε, σημασία. Γι' αυτό και θεωρώ ότι δεν είναι ε, δόκιμος ο όρος αυτός. Τρίτον, ο κύριος Γιόνκερ με συμπεριέλαβε στη διαδικασία. Με ρωτήσατε αν συμμετείχα. Ναι, συμμετείχα. Αν είχα μάλιστα εκφράσει αντιρρήσεις μου ως προς τις, τα προσόντα του υποψηφίου, δεν θα είχε καταλήξει η πρόταση αυτή στο Σώμα των Επιτρόπων. Αντίθετα όμως, εγώ είμαι βαθιά πεπισμένος για τις ικανότητες του ανδρός, γιατί τον γνωρίζω εδώ και 8 χρόνια. Καθημερινά συνεργαζόμαστε. Αν ήξερα την πρόθεση του κυρίου Ιταλιάνερ νωρίτερα. Και αν ήταν ένα θέμα το οποίο το ήξερε μόνο ο κύριος Ιταλιάνερ και μόνο ο κύριος Γιούγκερ και είχε υπάρξει μια διαρροή, τότε ναι, ενδεχομένως θα ε, μου είχαν ε, γεννηθεί και εμένα διάφορα ερωτηματικά. Όμως δεν υπήρξε κάτι τέτοιο, γι' αυτό και είμαι πάρα πολύ ικανοποιημένο από τη διαδικασία που ακολουθήθηκε. Σε πρώτη φάση η απόφαση αυτή βεβαίως αφορά τα προσόντα, τα ουσιώδη προσόντα του υποψηφίου, είναι όμως και μια πολιτική αποφάση. Διότι ο πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής χρειάζεται κατά την εκτέλεση των πολύ σημαντικών καθηκόντων του να έχει συνεργάτες που τους εμπιστεύεται προσωπικά, πολιτικά, διοικητικά Ακριβώς διότι είναι αναγκαίο οι άνθρωποι που τον περιβάλλουν, τον πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, να έχουν τα απαραίτητα προσόντα. Είπατε μάλιστα ότι ε, ενεργήσαμε περίπου σαν τον Τραμπ. Νομίζω ότι δεν ισχύει καθόλου αυτό. Στην Κομισιόν ακολουθούμε τελείως διαφορετικές διαδικασίες από την κυβέρνηση Τραμπ. Και αν θεωρείτε ότι στις απαντήσεις μας περιλαμβάνονται ψεύδι, παρακαλώ να μου πείτε σε ποια ακριβώς ερώτηση, σε ποια απάντηση, σε ποια σελίδα. Νομίζω ότι είναι απαράδεκτο να μας κατηγορείτε ότι χρησιμοποιούμε ψεύδι, γιατί κάθε άλλο παρά ψεύδι έχουμε χρησιμοποιήσει. Κύριος Στάς. Ευχαριστούμε κύριε Πρόεδρε. Κύριε Τιγκερ, μάλλον δεν καταλαβαίνετε, δεν συνειδητοποιείτε πόσο έχει βλαβεί η φήμη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Αυτά τα οποία μας λέτε δεν διαψεύδουν το ότι δεν έγιναν τα πράγματα με διαφάνεια. Θα μπορούσε να υπάρξει μια ανοιχτή διαδικασία, μια διαδικασία με διαφάνεια όπως προβλέπει το άρθρο 29 του καταστατικού εσείς διάλεξατε μια άλλη διαδικασία πρώτα πρώτα το 2015 είχε γίνει γνωστό ότι θα πάρει σύνταξη το 2018 την άνοιξη ο κύριος Σταλιάνερ. αυτό το ήξερε ο κύριος και ο κύριος Γιούγκερ εσείς με θα έπρεπε αρκετά νωρίς να έχετε ενημερωθεί σε σχέση με το τι θα γινόταν με τον κύριο Ταλιάνερ πριν τις 20 Φεβρουαρίου. Ο κύριος Μπράντι, σας αν δεν θεωρείτε ότι αυτό σημαίνει δυσπιστία προς το πρόσωπό σας, μα δεν θα έπρεπε να έχετε καλύτερη διαχείριση του προσωπικού και να είσαστε προετοιμασμένοι για τη διαδικασία αντικατάστασης έχοντας μάθει ότι ο κύριος Ιταλιάνε θα αποχωρούσε την άνοιξη του 18. Συμφωνείτε ή όχι, κύριε Τιγκερ, ότι η όλη διαδικασία για τον ορισμό του κυρίου Σελμάγερ ως η Γενικού Αματέα έγινε ούτως ώστε να πάρει αυτή την θέση και έτσι να είναι ο σίγουρος διάδοχος του κυρίου Ιταλιάν άμα την αποχώρησή του. Επίσης, επικαλεστήκατε το άρθρο 7 ε, για τη διαδικασία αυτή από πλευρά σας, που λέει τόσο, για, για το συμφέρον της υπηρεσίας και μας είπε η νομική υπηρεσία του Κοινοβουλίου ότι είναι δυνατόν ε, για το συμφέρον τη υπηρεσία κάποιο να αλλάξει καθήκοντα, να μετακινηθεί, αλλά μόνο όταν η κατάσταση είναι ιδιαίτερο σοβαρή, ε, και κατεπήγει αυτή η μεταβολή. Στις 21 Φεβρουαρίου τι ακριβώς συνέτρεχε από αυτές τις συνθήκες. Υπήρχε κάποιο γεγονός τόσο σπουδαίο, τόσο επίγον, δεν μπορούσατε να τα αναβάλλετε αυτά και 28 Δευτέρω Και 1η Μαρτίου να πάμε πάλι είχατε για την φυσιολογική διαδικασία αρκετό χρόνο. Τέσσερις εβδομάδες σε τρεις εβδομάδε έγινε προεδρής Γενικός Γραμματέα, άρα θα είχατε τον απαραίτητο χρόνο. Μπορούσατε να περιμένετε μέχρι την 1η Απριλίου, ε, να περιμένετε μέχρι την στέξη του κυρίου Τελειάνα. Μα τι κοπάδι είναι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Δεν αναλαμβάνουν το ρόλο τους γιατί έχουν ε, διατελέσει αξιωματούχοι που είναι πολύ σημαντικά καθήκοντα. Μα είναι δυνατόν κάτι να ολοκληρωθεί, κάτι να δεκυπηρεωθεί στο γόνατο μέσα σε 9 λεπτά, γιατί έτσι ε, απίτησε ο κύριος Γιούνκερ. Κύριε πίτρο. Ε, οπ, Herr Το αν ε, ο κύριος Γιούνκερ δεν με εμπιστεύεται, δεν είμαι εγώ ε, αυτός που μπορώ να το αξιολογήσω. Εγώ δεν θεωρώ ότι ε, δεν την χάνω της ε, εμπιστοσύνης του κυρίου ε, Όπως είπα, αν είχα εκφράσει αντιρρήσεις, δεν θα είχε προχωρήσει στην υποβολή αυτής της πρότασης. Τώρα, ως προς τον διορισμό έκπληξη που αναφέρατε, και τις, την παράκαμψη των διαδικασιών. Έχουμε απαντήσει σε αυτά. Τόσο στην περίπτωση του κυρίου Έμι Τσάλιβαν, όσο και στην, στην περίπτωση Κάθριν Ντέι και του κυρίου Ιταλιάνερ, η διαδικασία ήταν πάντοτε ίδια, χωρίς προκήρυξη. Και μάλιστα τότε, την άνοιξη του 2015, στο πλαίσιο της συνεδρίασης της Κομισιόν, ως Επίτροπος Ψηφιακής Οικονομίας είχα ενημερωθεί ότι η Κάτριν Ντέι επιθυμεί να συνταξιοδοτηθεί. Τότε λοιπόν έμαθα για τον διορισμό του κυρίου Ιταλιάνερ και συμφώνησα. Εσείς ε, δεν ξέρω τι ακριβώς εννοείτε ε, ως προς την ασφαλή θέση που αναφέρατε. Η θέση του Γενικού Γραμματέα είναι πολύ σημαντική, καθόλου ασφαλής όμως. Δεν είναι διαβίου μόνιμος. Κάθε επόμενη Κομισιόν, κάθε επόμενη ε, Ευρωπαϊκή Επιτροπή μπορεί να αλλάξει τον Γενικό Γραμματέα. Για απέτηση του κυρίου Γιούγκερ επίσης προς την ε, Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν μπορώ να κάνω λόγο. Ήρθε στο Σώμα των Επιτρόπων και μας εξήγησε γιατί πρέπει να κάνει δεκτή την αποχώρηση του κύριου Ιταλιάνερ και γιατί θεωρεί ότι ο κύριος Σέλμαερ είναι ο καταλληλότερος να τον διαδεχτεί χωρίς να υπάρξει καμία αντίρρηση. Μιλώντας λοιπόν για πρώην πρωθυπουργούς και το ειδικό πολιτικό βάρος που τους χαρακτηρίζει είναι προφανές ότι κάθε επίτροπος, αν διαφωνούσε, θα μπορούσε να είχε εκφράσει τις αντιρρήσεις του. Το γεγονός ότι κάτι τέτοιο δεν συνέβη, δεν σημαίνει βεβαίως ότι ήρθε, να ήρθε, ε, ότι ήρθε ο κύριος Γιούγκερ και επέβαλε την ε, θέλησή του. Πρόεδρος, προφανώς η διαδικασία επιλογής ε, και διορισμού Γενικού Γραμματέα βρισκόταν στην, στην ε, ημερήσια διάταξη εκείνης της συνεδρίασης. Ο κύριος Ντεγιόν. Ευχαριστώ Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε. Θα ήθελα καταρχάς να γνωρίζω Ποια είναι η αντίδρασή σα σε σχέση με μια δήλωση του κυρίου Σελμάιρ που είπε ότι ήδη πριν τα Χριστούγεννα γνώριζε τι θα συνέβαινε. Άρα είχε ενημερωθεί προσωπικά και εγκαίρως από τον κύριο Γιούνκερ ότι επρόκειτο να γίνει αυτή η αλλαγή. Και γνώριζε ήδη από τότε ότι ο κύριος Γιούγκερ θεωρούσε τον ίδιο τον κύριο Σελμάιρο τον πλέον κατάλληλο να δεδεχθεί τον κύριο Ιταλιάνερ. Εκπρόσωπο Ευρωπαϊκή Επιτροπή το έχει πει αυτό. Εσεί τι έχετε να πείτε γι' αυτό. Πρώτον αυτό. Δεύτερον. Λέτε ότι καμία δυσαρέσκεια δεν ακούστηκε στα πλαίσια της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Πολύ ωραίο αυτό. Εγώ θα έλεγα όμως ότι ένα σύλλογος γανουβό δημοκρασί εξέφρασε πραγματικά ανησυχίες και δυσαρέσκεια για την όλη διαδικασία και ζήτησε να ακολουθηθεί μια ανοιχτή διαδικασία και γενικότερα να ακολουθούνται πολύ πιο διαφανείς διαδικασίες. Για πρόβλημα λοιπόν δεν έγινε κάτι τέτοιο. Για ποιο λόγο δεν αναθεώρησε επίσης την όλη αποφασή της Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Και τέλος, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μας λέτε ότι δεν συμφωνεί με τα όσα εμείς προσάπτουμε. Λέτε ότι είστε ένα πολιτικό όμως όργανο παίρνετε μια απόφαση και προκαλεί τεράστια αναστάτωση αυτή στην κοινή γνώμη και στους δημοσιογράφους. Αναφερθήκαμε εμεί στη στρατηγική που ακολουθεί για τα μέσα μαζική ενημέρωση και εσεί αναφερθήκατε πολύ απλά σε μία συνέντευξη τύπου. Μα καταλαβαίνετε ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό εσεί να γίνεστε αποδέκτη πραγματικά και να είστε σε θέση να αφουγκράζεστε τη δυσαρέσκεια που εκφράζεται από δημοσιογράφου και γενικότερα από την κοινή γνώμη και τη δυσαρέσκεια αυτή να λαμβάνετε πολύ σοβαρά υπόψη σα και τη συνεχεία να δίνετε και τι κατάλληλε απαντήσει. Έχω την εντύπωση ότι αντιμετωπίσετε την κοινή γνώμη και εν γέννη του δημοσιογράφου αλλά και του ευρωβουλευτέ σαν μικρά παιδιά. Ουσιαστικά προσπαθήσετε να παρακάμψετε εντελώ οποιαδήποτε διαδικασία λογοδοσία. Μπορούμε να πούμε λοιπόν ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι ένα θεσμικό όργανο που έχει χάσει κάθε επαφή με την κοινωνία Νομίζω ότι αληθεύει αυτό και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρέπει έστω και τελευταία στιγμή να δείξει ότι νοιάζεται για τι ανησυχίε των πολιτών. Ευχαριστώ. Το ότι έγινε προκήρυξη της, ε, της θέσης του Γενικού Γραμματέα εδώ δεν το αμφισβητώ βεβαίως, όμως μην ξεχνάτε ότι εδώ υπάρχει ε, υπάρχουν πολιτικές ομάδες. Ποιο θα είναι γενικός γραμματέας, αποφασίζεται εκεί ποιο είναι αναπληρωτή γενικό γραμματέας. Γι' αυτό και η συγκρισιμότητα μεταξύ Κομισιών και Κοινοβουλίου είναι περιορισμένη. Δεύτερον, τα δελτία τύπου ε, που έχουμε εκδώσει ε, τα λένε ήδη όλα. Ο κύριος Σελμάιερ ήταν διευθυντής του γραφείου και συνεργάτης του ε, κύριου Γιόνκερ. Ήταν βεβαίως ενήμερος για το γεγονός ότι ο κύριος Ιταλιάνερ δεν ήθελε να εξαντλήσει τη θητεία της Κομισιόν στη θέση του Γενικού Γραμματέα. Όμως, νομίζω ότι και υπάρχουν ε, τεκμήρια γι' αυτό, Έως και τον Φεβρουάριο ο κύριος Γιούγκερ προσπαθούσε να πείσει τον κύριο Ιταλιάνερ να παραμείνει στη θέση του. Υπάρχουν τεκμήρια, ξαναλέω. Εμείς, εγώ προσωπικά και το επιτολείο μου συνεργαστήκαμε πολύ στενά ε, με τον ε, κύριο Ιταλιάνερ και είχαμε την ευκαιρία πολλές φορές να το εκφράσουμε αυτήν μας την επιθυμία. Θα συζητήσω το θέμα αυτό και μετά συνδικάτα, τα οποία και θα συναντήσω μετά την ε, τωρινή μας, την συνεδρίασή μας, τη συζήτησή μας αυτή. Είπατε να μην κρυβόμαστε πίσω από νομικούς κανόνες. Μα με συγχωρείτε πάρα πολύ. Εγώ απάντησα στις 134 ερωτήσεις σας. Ακριβώς διότι θεωρώ το θέμα πολύ σημαντικό. Αλλά τα ερωτήματά σας είναι νομικής φύσης. Γι' αυτό και απαντώ με βάση τις νομικές μου γνώσεις και με βάση την νομική μου αντίληψη. Αν θέλατε να με ρωτήσετε για τα συναισθήματά μου ή για τον καιρό, θα σας έδινα άλλες απαντήσεις. Αλλά οι δικές σας ερωτήσεις ήταν νομικής φύσης και αφορούσαν το κατά πόσο τηρήθηκαν οι κανόνες δικαίου που εσείς έχετε θεσπίσει στον κανονισμό του προσωπικού. Επίσης, εγώ ήμουν 26 χρόνια βουλευτής στη Βάδε Βιτεμβέργη. Είμαι κοινοβουλευτικός άνδρας λοιπόν. Έχω εμπειρία κοινοβουλευτική σε τοπικό, περιφερειακό και εθνικό επίπεδο. Πολύ περισσότερο ε, η πολύ περισσότερη και πολύ μεγαλύτερη είναι η κοινοβουλευτική μου εμπειρία παρά εκείνη που έχω στην εκτελεστική εξουσία. Γι' αυτό και σε καμία περίπτωση δεν θέλω να δημιουργήσω την εικόνα και την αίσθηση σε εσά ότι σας αντιλαμβάνομαι ή σας συμπεριφέρομαι σαν παιδάκια. Θεωρώ πολύ σημαντικά αυτά τα θέματα, γι' αυτό και ε, βρίσκομαι εδώ και συζητώ μαζί σας. Δεν νομίζω ότι μπορεί κανείς να με κατηγορήσει ότι είμαι ένας άνθρωπος απογειωμένος, αποκομμένος από την πραγματικότητα. Την προηγούμενη εβδομάδα ήμουνα στην Πολωνία. Συναντώ ανθρώπους καθημερινούς, απλούς πολίτες. Μιλώ μαζί τους για τις ανησυχίες τους, για τους προβληματισμούς τους, για τους φόβους τους. Γι' αυτό σας παρακαλώ μην τροφοδοτούμε τους λαϊκιστές, που έξω από εδώ, από τις Βρυξέλλες, ισχυρίζονται ότι είμαστε απογειωμένοι και αποκομμένοι από την πραγματικότητα. Δεν ισχύει αυτό. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Άκουσα τον Επίτροπο, άκουσα τα όσα είπε. Μας είπε για την πολιτική αυτή φύση του διορισμού Σελμάιερ. Τον ήθελε πραγματικά ο Γιούνκερ, τον Σελμάιερ στη θέση αυτή το ΕΛΚ επίσης τον ήθελε, άρα είναι μία απόφαση που ελήφθη σε πολύ ψηλό επίπεδο και στα πλαίσια του ΕΛΚ προκειμένου να μπορούμε να έχουμε ως υψηλό βαθμό ή τον πιο υψηλό βαθμό πλέον δημόσιο υπάλληλο στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή έναν άνθρωπο ο οποίος θα ήταν ε, από πολιτικής πλευράς άξιος εμπιστοσύνης, τουλάχιστον όσον αφορά το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα. Εγώ όπως και πολλοί άλλοι θεωρούμε ότι δεν θα έπρεπε να είχε ακολουθηθεί μια τέτοια προσέγγιση σε αυτό το διορισμό, μια πολιτική δηλαδή προσέγγιση. Ξέρω ότι αυτή τη στιγμή υφίστανται κάποια νομικά ζητήματα, γιατί δεν καταλάβαμε τελικά πάρα πολύ καλά αν έγινε ή όχι, πώς έγινε η προκήρυξη της θέσης αυτής. και νομίζω τελικά ότι θα πρέπει να είχαμε δει διαφορετικά αποτελέσματα από ό,τι είδαμε τελικά για τη δημοσίευση αυτή, καθότι δεν υπήρχαν και, και πολλοί υποψήφοι. Πρέπει λοιπόν να δούμε ποιοι είναι οι κανόνες όσον αφορά τον διορισμό, αν ακολουθήθηκαν οι κανόνες αυτοί. Εδώ υπάρχει μια διάσταση απόψεων στο Κοινοβούλιο. Μιλάμε πάντως, θεωρώ, για έναν διορισμό πολιτικό. Επομένως, θα πρέπει η Επιτροπή Γιούνκερ να δεσμευτεί ρητά ότι εφόσον έχει ακολουθηθεί τελικά μια πολιτική διαδικασία, θα πρέπει ο άνθρωπος αυτός να απομακρυνθεί και να ακολουθηθεί μια άλλη διαδικασία, η οποία να συνάδει τελικά και με τις προσδοκίες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Καθότι λοιπόν ήταν ένας ηθελημένος από τον Γιούγκερ διορισμός αυτός, και καθότι μπορούμε να πούμε τελικά ότι ο Γιούνκερ είναι ο τελικό υπεύθυνο για το διορισμό αυτό, προφανώ έδωσαν την έγκρισή του στη ε, συνεχεία και οι επίτροποι, αλλά ο πλέον υπεύθυνο είναι ο Γιούνκερ, μην το ξεχνάμε αυτό. Ε, Μήπω δεν θα έπρεπε να ακούσουμε και τον Γιούνκερ, καθώ είναι ο πλέον υπεύθυνο παράγοντα, αν θέλετε, στην όλη αυτή η ε, ιστορία. Νομίζω ότι θα ήταν σημαντικό και πρέπει να το πούνε και οι υπόλοιποι συνάδελφοι αυτό, και αυτοί συμφωνούν, να ακούσουμε και τον ίδιο τον κύριο Γιούνκερ σε αυτή την επιτροπή. Επίτροπε, έχετε το λόγο. Die letzte Frage ist eine Frage an Sie selbst und an Ihr Präsidium. Η τελευταία ερώτηση. Ε, λέει ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ό,τι ζητάτε σας το λέει. Ναι, η πόρτα είναι ανοιχτή. Αν θέλετε, να το και στο Στασβούργο. Να τα συζητήσουμε όσο θέλετε, όσο έχουμε συμφωνήσει. Μιλήσατε για το τέλος της ε, θητείας της Κομισιόν Γιόγκερ. Έχουμε άλλους 19 μήνες. Σχεδόν το 1 τρίτο, δηλαδή. Δεν βρισκόμαστε δηλαδή στο τέλος της θητείας. Στο μέσον βρισκόμαστε. Ίσως από το φετινό Πάσχα έως του χρόνου το Πάσχα μάλιστα είναι και η σημαντικότερη περίοδος της θητείας μας. Γι' αυτό και είναι πάρα πολύ σημαντικό όταν κάποιος υψηλόβαθμος αξιωματούχος θέλει να αποχωρήσει και δεν πείθεται να παραμείνει, χρειάζεται να καλυφθεί η θέση αυτή άμεσα προκειμένου να εξασφαλιστεί η δυνατότητα δράσης της Κομισιόν. Αν εδώ είχαμε περάσει 4 ή 8 εβδομάδες χωρίς γενικό γραμματέα και κάτι πήγαινε στραβά, δικαίως θα μας λέγατε ότι δεν μπορούμε να δράσουμε και να ανταποκριθούμε στις υποχρεώσεις μας. Γι' αυτό, άμα δείτε το χρονοδιάγραμμα ε, της νομοθετικής διαδικασίας, των τριμερών διαλόγων, της προετοιμασίας του προ, για όλους αυτούς τους λόγους, εγώ σας λέω ότι χαίρομαι που η θέση αυτή κατέστη δυνατό να καλυφθεί με έναν ικανό υποψήφιο άμεσα. Εγώ δεν έχω ρωτήσει ποτέ τον κύριο Σελμαρέ αν είναι κομματικό μέλος. Διάβασα στα μέσα μαζικής ενημέρωσης ότι δεν ανήκει στο κόμμα μου. Το σημειώνω αυτό. Αν κάποια στιγμή λάβω κάποιο, κάποια αίτηση προσχώρησης, βεβαίως θα σας το κοινοποιήσω και εσάς. Εγώ γνωρίζω ότι ο άνθρωπος αυτός δεν είναι μέλος του Τσεντεού και του Τσέσου. Το γεγονός ότι εγώ ανήκω στο ΕΛΚ, όπως και ο πρόεδρος Γιούγκερ, ε, να με συγχωρείτε. Εγώ είμαι μέλος του Τσεντεού εδώ και 4, 40 χρόνια και δεν έχω σκοπό να αποχωρήσω. Σας το λέω. Όμως, υπερκομματικά και αντικειμενικά εκπληρώνω τα καθήκοντά μου. Γι' αυτό και λέω σε εσάς ότι έχω πρόθεση και θέλω να μετεξελίξω και να εκπληρώνω τα καθήκοντά μου αντικειμενικά και χωρίς κομματικές παροπίδες. Και νομίζω ότι αυτό είναι ένα χαρακτηριστικό και του κυρίου Γιούγκερ. Και νομίζω ότι είναι και ένα χαρακτηριστικό που ε, διακρίνει πολλά μέλη του ΕΛΚ που βρέθηκαν σε υψηλόβαθμες θέσεις εντός των ευρωπαϊκών θεσμικών οργάνων. Γιούγκερ, Έτιγκερ, Τίμερμανς, όχι μόνο ε, εμείς οι τρεις, ήταν και ο Τίμερμανς ήταν ε, ε, ενήμερος, υποστήριξε την ε, συγκεκριμένη ε, πρόταση, όχι μόλις την Τετάρτη το απόγευμα, αλλά από την Τρίτη το βράδυ και ο Τίμερμανς είναι ένας πολύ ευφυής άνδρας, τον οποίο δεν μπορεί κανείς εύκολα να παραπλανήσει και ανήκει στην πολιτική ομάδα των σοσιαλιστών από τις κάτω χώρες. Αν επρόκειτο για πολιτικό διορισμό, εγώ θα έλεγα ότι πρόκειται για έναν ε, διορισμό βάσει ικανοτήτων και προσόντων που βεβαίως έχει πολιτική σημασία και που θεωρώ ότι δεν ήταν εσφαλμένη. Το αν ήταν ορθή η απόφαση αυτή μπορεί να το αποδείξει η Κομισιόν και ο νέος Γενικός Γραμματέας τους επόμενους 19 μήνες. Βεβαίως, ελέγχεται. Τους επόμενους 19 μήνες θα διαπιστώσετε αν θα διαψευστώ ή αν θα επιβεβαιωθώ στην εκτίμησή μου αυτήν που σας εκφράζω αυτή τη στιγμή. Αν και εγώ θεωρώ ότι δεν θα διαψευστώ. Επίτροπε, βρισκόμαστε εδώ πέρα για να καταλάβουμε λίγο την μπαρόκ αυτή διαδικασία που ακολουθήθηκε προκειμένου να εκτοξευθεί στη θέση του Γενικού Γραμματέα ο κύριος Σελμάιρο, που ήταν πρώην επικεφαλής του γραφείου του κυρίου Γιούνκερ. Διακριτική μεταχείριση, προνομιακή μεταχείριση, εντελώς αδιαφανής, που πραγματικά παραβαίνει όλους τους κανόνες που θα πρέπει να ισχύουν προκειμένου να έχουμε μια αξιοκρατική Ευρωπαϊκή Επιτροπή και Ευρωπαϊκή Δημόσια Διοίκηση. Θα πρέπει να μας ξεκαθαρίσετε ότι όντως ακολουθήθηκε το άρθρο 2 της Ευρωπαϊκής Ένωσης που λέει ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση βασίζεται στο κράτος δικαίου. Ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ακολούθησε όντω τη συμφωνία τη Οργανική του 2016 για το 7ο θετήν. 3. Ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παράλληλα έχει ένα μητρό διαφάνεια και το επιβάλλει σε όλου του οργανισμού και σε όλα τα άτομα τα οποία ανεξάρτητα συμμετέχουν ε, στην επεξεργασία και εφαρμογή των πολιτικών τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Εφόσον αυτό το επιβάλλουμε στου άλλου, πρέπει να το επιβάλλουμε και σε εμά του ίδιου. Θα θέλαμε λοιπόν να καταλάβουμε για ποιο λόγο ένα μέλος του γραφείου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής γίνεται ξαφνικά Γενικός Γραμματέας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής χωρίς να έχει αναλάβει ποτέ τη θέση ε, διευθυντή, χωρίς να είναι ποτέ επικεφαλής ε, γενικής διεύθυνσης και χωρίς να έχει προκηρυχθεί καν η θέση αυτή. Υπήρχαν πάρα πολλοί άλλοι αξιόλογοι και ικανότατοι ε, υπάλληλοι της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που δεν είχαν τη δυνατότητα να προχωρήσουν τόσο γρήγορα όσο ο κύριος Σελμάιερ. Στις αρχές του 2017 ο κύριος Σελμάιερ είχε πει ότι με τίποτα δεν θα αποδεχόταν τέτοιε πρακτικέ στα πλαίσια τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Μα στην πράξη είδαμε ότι όλα αυτά συμβαίνουν όχι μόνο με τη δική του υπόθεση, αλλά ακόμα και με την υπόθεση του κυρίου Μπαρόζο, ο οποίο πήγε πάρα πολύ εύκολα μετά στην Goldman Sachs, αφού του τελείωσε η θητεία του στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Και έπειτα έρχεται ο κύριο Γιούνκερ, ο οποίο πραγματικά δεν δείχνει καμία απολύτως ακεραιότητα όσον αφορά το ζήτημα αυτό. Αντίθετα, δείχνει μια ιδιαίτερα ευνοϊκή στάση απέναντι στον κύριο Σερμάγερ και αυτό φάνηκε και από τη στάση που κρατούσε απέναντι στο ίδιο το Ευρωπαϊκό το Κοινοβούλιο. Α μην ξεχνάμε βέβαια ότι εδώ και στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο τέτοια φαινόμενα είχαμε με τον πρώην πρόεδρο, τον κύριο Σούλτ, ο οποίο προτού αποχωρήσει από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο φρόντισε να τακτοποιήσει σε πάρα πολύ καλέ θέσει διάφορου ε, δικούς του υφισταμένους. Μας λέτε ότι όλα αυτά αιτιολογούνται τώρα από το ανώτο συμφέρον της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Υπηρεσίας. Αυτό είναι το νεοδόγμα το οποίο θα προωθεί πλέον η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για να δικαιολογήσει τα κακό κείμενα. Κύριε Επίτροπε. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή με τη σύμφωνη γνώμη του Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου αποφάσισε ότι μετά την ολοκλήρωση μιας θητείας στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και την ανάληψη καθηκόντων ε, εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, θα πρέπει να ε, ανέρχεται σε τουλάχιστον δύο χρόνια και για τον πρόεδρο της Κομισιόν τρία χρόνια. Εγώ δεν γνωρίζω αυτή τη στιγμή κανένα κράτος μέλος, ούτε και κανένα κράτος στον κόσμο, να υπάρχει μια τέτοια διαδικασία, μια τέτοια περίοδος ε, όπου κανείς δεν επιτρέπεται μετά την ανάληψη δημόσιων καθηκόντων να αναλάβει ε, άλλη θέση. Νεποτισμός και αναξιοκρατία. Εγώ δεν ξέρω και ε, ε, ο, πρέπει να σας πω ότι ο κύριος Σέλμαϊρ δεν είναι συγγενής του κυρίου ε, Γιούγκερ. Βεβαίως είναι εμπιστός του και είναι προφανές. Ένας πρόεδρος πρέπει να έχει εμπιστοσύνη στον υφιστάμενό του και μάλιστα σε έναν τόσο υψηλό βαθμό υφιστάμενό του. Αυτό είναι δεδομένο, απαραίτητο, λογικό και αναγκαίο. Δεδομένου λοιπόν ότι ο κυριος σελμαιρ Σελμάιερ ήταν AD15 βαθμός και εξακολουθεί να έχει βαθμό AD15 η αλλαγή του στην θέση του Γενικού Γραμματέα είναι και νόμιμη και εύλογη. Τα επιτελεία και τα γραφεία στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή διαδραματίζουν πολύ σημαντικό ρόλο. Ένας επικεφαλής γραφείου και επιτελείου έχει σε ορισμένες περιπτώσεις και μάλιστα στις περισσότερες περιπτώσεις περισσότερα ε, καθήκοντα, περισσότερες υποχρεώσεις από οποιονδήποτε γενικό διευθυντή. Είναι λοιπόν σωστό ότι αν το μοναδικό κριτήριο ήταν η ηλικία ή τα χρόνια υπηρεσίας, βεβαίως η προαγωγή του κυρίου Σελμάιρ ήταν πολύ ταχεία. Αλλά σας το λέω ξεκάθαρα γιατί εγώ έχω έρθει αντιμέτωπος πολλές φορές με αυτό το ερώτημα. Γιατί θα πρέπει να προκρίνονται πάντοτε ε, εκείνοι που έχουν τη μεγαλύτερη ηλικία ή τη μεγαλύτερη ε, υπηρεσιακή ηλικία, αν το θέλετε έτσι. Όχι. Θεωρώ ότι πρέπει να είμαστε σε θέση, όχι μόνο μέσω των ευρωεκλογών, ε, αλλά σε όλα τα επίπεδα, να έχουμε τη δυνατότητα να έχουμε και πρωθυπουργό ο οποίο είναι 31 ετών. Ε, λοιπόν θα πρέπει να μπορούμε να έχουμε και την εμπιστοσύνη, εμπιστοσύνη σε έναν 47χρονο άνδρα ότι μπορεί να εκτελέσει τα καθήκοντά του. Από αυτή την άποψη λοιπόν πριν από πολλά χρόνια υπήρξε στην κυρία, ε, στην, στην, στο επιτελείο της ε, κυρίας Δαμανάκη ε, μια τμήματαρχη, η οποία έγινε γενική διευθύντρια και ε, ήταν διευθύντρια του, του, ε, του γραφείου της κυρίας Δαμανάκη, η οποία πράγματι παρέμεινε στη θέση της. Ίσως χωρίς ποσόστοση δεν θα είχαμε, καταλήξουμε, δεν θα είχαμε καταλήξει σε αυτή την απόφαση. Αν όμως θεωρούμε ότι είναι σοβαρό θέμα η ποσόστοση γυναικών, τότε πρέπει να επιμένουμε και να εμένουμε σε αυτήν την ε, διαδικασία επιλογής προσωπικού. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, ε, Επίτροπε. Θέλω να σας πω ότι φυσικά η ίση μεταχείριση των υπαλλήλων είναι επίσης πολύ σημαντική. Γι' αυτό και ε, καταλαβαίνω γιατί δημιουργήθηκε αυτή η ταραχή στις υπηρεσίες της ε, Κομισιόν. Και βεβαίως ε, σε αυτό απαντά και το θέμα της ποσότητας των γυναικών. Ακριβώς γιατί συνδέεται με τις ίσες ευκαιρίες για όλους τους ανθρώπους. Λοιπόν, συνεχίζουμε τώρα με τους, ο, τις παρεμβάσεις από τις πολιτικές ομάδες. Ο κ. Χαΐζης έχει το λόγο. Thank you, Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Πρώτα απ' όλα επίτροπε, ας ανατρέξουμε στην απαντησή της ερωτήσεως 32 όπω και τα είπε προηγουμένω και σα ερώτησε ο κύριο Ελισάντρου για το κατά πόσο εσεί και ο κύριο Γιούγκερ τα γνωρίσατε και στην απάντηση είπατε ότι το 2015 ήξερε για την επικείμενη συνταξιοδότηση του κύριου Ιταλιάνερ και ότι αρχάς το 2018 υπήρξε άποψη ότι θα τηρούσε την απόφασή του και τώρα στις αρχές του 2018 εσείς πώς μπορείτε να υποστηρίξετε αυτό το πειράζει στην απαντησή σας ότι δηλαδή αρχάς του 2018 ο κύριος Ταλιάνο επεβεβαίωσε ότι θα ε, τηρήσει, θα υλοποιήσει την απόφασή του. Αυτό ποιος το επιβεβαίωσε. Γιατί εσείς θα πρέπει να έχετε την αίσθηση ότι σας ξεγέλασαν. Σας πετάξαν εδώ μέσω της Επιτροπής μας για να υπερασπίσετε ε, όλα αυτά τα οποία έγιναν. Αφού είστε ο υπεύθυνο για το προσωπικό, γιατί δεν ξέρετε τίποτα. Νομίζω ότι είναι σημαντικό να παίζει το φως για το ποιο και πότε ήξερε τι. Στην απάντησή σας όσον αφορά το ερώτημα 19, εκεί που λέτε ότι δεν υπήρχε νομική υποχρέωση για το κατά να υπάρξουν περισσότεροι υποψήφοι και ότι ένας αρκούσε. Δεν πρόκειται για ανώνυμη εταιρεία. Πρόκειται για ένα πάρα πολύ θεσμικό, διεθνή οργανισμό που έχει υποχρεώσεις ε, αποδόσεως και αναλήψεως ευθυνών και ότι θα πρέπει η κάθε απόφαση του οργανισμού να διακρίνεται από νομιμότητα. Και υπάρχει, δεν συμφωνείτε, πολιτική υποχρέωση από πλευρά διαφάνεια όλα αυτά να γίνουν έτσι, ούτω ώστε να υπάρχουν περισσότεροι υποψήφοι. Και η τελευταία ερώτηση μα ε, μιλήσατε για την επόμενη επιτροπή, τον επόμενο πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Τι πιστεύετε Όχι, όχι, όχι, δεν τον επικοινωνώ προσωπικά, γιατί είναι ικανότατο. Είναι κάποιο που έχει τεραστία εμπειρία στο management και στη διαχείριση, αλλά σε σχέση με κάτι που έπρεπε προηγουμένω σε συνάδελφο, ότι κατά κάποιο τρόπο η θέση του κ. Σελμάγερ δεν θα υπάρχει με το που θα φύγει ο κύριο ε, Γιούνκερ. Και ο νέος, και ο γραμματέας, και ο νέος πρόεδρος της Επιτροπής πρόκειται να ορίσει κάποιον άλλον. Ισχύει αυτό. Επίτροπε, έχετε τον λόγο λοιπόν. Μετά από πολλέ συζητήσεις που έχω κάνει, θεωρώ δεδομένο ότι ο κύριος Γιούνκερ την άνοιξη του 2015 μετά την ε, αποχώρηση της κυρίας Ντέι και εφόσον είχε προετοιμαστεί φάκελος όπως ψηφίταν από την κυρία Γκοργίεβα την προκάτεχό μου, κατέληξε στην, στο συμπέρασμα ότι πρέπει να βρεθεί μια λύση για τη διαδοχή της κυρίας Ντέι. Έλαβε λοιπόν την σύμφωνη γνώμη του κυρίου Ιταλιάνερ, προκειμένου να ολοκληρωθεί αυτή η μετάταξη από την ε, ε DG.com στη θέση του Γενικού Γραμματέα, επισημένοντας βεβαίως τότε ο κύριος Ιταλιάνερ ότι τον Μάρτιο του 2018, τρία χρόνια αργότερα δηλαδή, επρόκειτο είχε ε, πρόθεση να αποχωρήσει. Οι δύο άντρες λοιπόν παρέμειναν σε επαφή και ο κύριος Γιόγκερ προσπάθησε επανειλημμένος στα τέλη του 2017 και στις αρχές του 2018 να ε, πείσει τον κύριο Ιταλιάνερ να παραμείνει στη θέση του έστω και για λίγους μήνες. Προσπάθησε να τον πείσει. Δεν τα κατάφερε. Και όταν πια ήταν σαφές ότι ο κύριος Ιταλιάνερ ήταν αποφασισμένος να συνταξιοδοτηθεί και να αποχωρήσει, αποφάσισε ότι η θέση του Γενικού Γραμματέα πρέπει να καλυφθεί άμεσα. Και γι' αυτό το σκοπό ενημέρωσε εμένα και τον συνάδελφο Τίμερμανς, όπως είχε υποχρέωση από τον κανονισμό να κάνει. Εμείς πάντοτε στην, ε, για την κάλυψη θέσεων θέλουμε να έχουμε πολλούς υποψήφιους. Χωρίς αυτό να σημαίνει ότι μπορούμε να εγγυηθούμε ότι κάθε θέση θα πρέπει, για την κάλυψη κάθε θέση, θα πρέπει να έχουν ε, υποβληθεί πολυάριθμες υποψηφιότητες. Αν μάλιστα υπάρχει υποψήφιος ο οποίος εκπληρώνει όλες τις προϋποθέσεις, θα ήταν άδικο απέναντι στον υποψήφιο αυτό να κυρώσει κανείς αυτήν την, ε, τη διαδικασία που μπορεί να ακολουθηθεί και να προχωρήσει σε προκήρυξη. Στις περιπτώσεις λοιπόν όπου υπάρχει ένας υποψήφιος ο οποίος με βάση την εκτίμηση του κυρίου Γιούγκερ, του κυρίου Τίμερμαντς και τη δική μου θεωρείται ότι είναι ότι έχει τις ε, ικανότητες, τότε φυσικά και πρέπει και καλά κάναμε, ε, προχωρήσαμε στον διορισμό του. Και έτσι καταλήξαμε στον διορισμό του κυρίου Σέλμαια. Βεβαίως, το ότι λογοδοτούμε ως Κομισιόν απέναντι σε εσά, απέναντι στο Συμβούλιο, απέναντι στο Ελεκτικό Συνέδριο, απέναντι φυσικά στην κοινή γνώμη, το δέχομαι απολύτως Επίσης, συμφωνώ μαζί σας ότι πρέπει πάντοτε να τηρείτε πλήρως η ισχύουσα νομοθεσία. Για το θέμα το ότι ο κύριος Σελμάιερ κατέκτησε μια ασφαλή θέση, έχω ήδη απαντήσει. Κανένας γενικός γραμματέας δεν είναι ισόβιος. Αυτό, αν αυτός ήταν ο σκοπός, του κύριου Γιούγκερ θα μπορούσε να είχε μεταθέσει τον κύριο Σελμάιερ σε θέση γενικού διευθυντή, για παράδειγμα. Ακριβώς διότι ο γενικός γραμματέας πρέπει πάντοτε να τη χάνει της εμπιστοσύνης των προϊσταμένων του και συγκεκριμένα του Προέδρου της Κομισιόν. Και αυτό με δεδομένο ότι θα έχουμε μια νέα Κομισιόν στα τέλη του 2019 επιτείνει ακόμα περισσότερο αυτή τη διάσταση. Κάθε υψηλόβαθμος αξιωματούχος της Κομισιόν ε, δεν, ε, κανένας μάλλον δεν είναι ισόβιος και αυτό είναι και θετικό. Ευχαριστώ Πρόεδρε, να ευχαριστήσω και τον Επίτροπο ιδίω για τις απαντήσεις του. Έφτασαν λίγο καθυστερημένα βέβαια, αλλά μας εξηγήσετε για ποιο λόγο φτάσανε με τέτοια καθυστέρηση. Να μας πείτε όμως και αν ενεπλάκει ο κύριος Σελμάιερ στη σύνταξη των απαντήσεων που υποβάλαμε εμείς. Μας είπατε επίσης ότι όσον σας αφορά ακολουθήθηκαν όλοι οι κανόνες, ότι όλα ήταν νομότυπα. Βέβαια πρέπει να αποδεχθούμε τις δηλώσεις σας, αλλά βέβαια πρέπει να πούμε ότι ε, τα πράγματα δεν φαίνονται πάρα πολύ θετικά ή τουλάχιστον φαίνεται να υπάρχει ένα πρόβλημα ως προς την αντίληψη της νομιμότητας της όλης διαδικασίας. Το είπε και ο κύριος και η κυρία Γιάννα Σέντερ πότε πραγματικά τελικά μαθεύτηκε ότι θα αποχωρούσε ο κύριο Ιταλιάντερ. Εσεί μα δώσατε κάποιε απαντήσει, αλλά νομίζω ότι θα υποβληθούν και περισσότερε ερωτήσει. Θα θέλαμε λοιπόν ή δυνατόν να μα δώσετε και κάποιε περισσότερε πληροφορίε και πέρα από τη σημερινή συνεδρίαση. Να κάνω τώρα μια πιο συγκεκριμένη ερώτηση όσον αφορά το μέλλον. Είναι πάρα πολύ σημαντικό εμεί να καταλάβουμε πώ θα εξελιχθούν τα πράγματα, να καταφέρουμε δηλαδή να διασφαλίσουμε ότι δεν πρόκειται κάτι τέτοιο, δεν πρόκειται κάτι τέτοιο να επανληφθεί στο μέλλον. Θα πρέπει στο μέλλον κάθε σχετική διαδικασία ήταν απόλυτα διαφανή επομένω. με όλα αυτά τα οποία συνέβησαν όπω συνέβησαν. Μπορείτε τώρα εκ των υστέρων να μα πείτε ότι θα μπορούσαν τα πράγματα να γίνονται κάπω διαφορετικά ή αν μη τι άλλο θα καταβάλλετε κάθε δυνατή προσπάθεια προκειμένου να διασφαλίσετε ότι στο μέλλον η διαδικασία θα είναι πιο διαφανή και ότι δεν πρόκειται τα ίδια λάθη να επαληθούν και στο μέλλον. Ο επίτροπο. Σα ευχαριστώ για την ε, πολύ ουσιαστική αυτή η ερώτηση. Όταν λάβαμε τον κατάλογο των ερωτημάτων, συζήτησα άμεσα με τον Διευθυντή Ανθρώπινων Πόρων, που είναι εδώ μαζί μου, και τον Διευθυντή του Γραφείου μου, και αναλύσαμε τις ερωτήσεις που μας αποστήλατε. Και ζητήσαμε να, συνταχθούν, να συνταχθεί ένα σχέδιο απαντήσεων στις ερωτήσεις αυτές. Στη συνέχεια στραφήκαμε προς την νομική υπηρεσία που ε, μας παρέχει συμβουλές όσον αφορά την εφαρμογή του κανονισμού προσωπικού. Στραφήκαμε και στον εκπρόσωπο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής προκειμένου να μας ενημερώσει σχετικά με υποψίες ή απόψεις που έχουν εκφραστεί στον ευρωπαϊκό τύπο. Συζητήσαμε με το επιτελείο του Προέδρου, με τον ίδιο τον Πρόεδρο και στα ερωτήματα που αφορούν προσωπικά τον κύριο Σελμάιερ, πότε ήξερε τι, συζητήσαμε τα θέματα αυτά προσωπικά με τον ίδιο. Μα πώς αλλιώς θα μπορούσαμε άλλωστε να απαντήσουμε αν δεν ε, παίρναμε την προσωπική του θέση, την προσωπική του άποψη. Πάντως υπεύθυνο για την ε, απάντηση των ε, ερωτήσεων δεν ήταν ο κ. Σελιμάιερ, ήμουν εγώ προσωπικά και όποτε εγώ δεν μπορούσα υπεύθυνο ήταν ο υπεύθυνο ο διευθυντής του γραφείου μου. Εγώ, όπως είπα, μπορώ να συζητήσω μαζί σας και διμερώς και στο επίπεδο συνεδρίασης πολιτικής ομάδας, είτε και εδώ στην Επιτροπή Κοντ και να μπούμε σε ακόμα μεγαλύτερο βάθος. Δεν θα αποφύγουμε, ούτε θα προσπαθήσουμε να αποφύγουμε τα ερωτήματά σας. Αντίθετα, θέλουμε να ενισχύσουμε την εμπιστοσύνη του Κοινοβουλίου προς την Κομισιόν και να εμβαθύνουμε τη συνεργασία μας. Για το ερώτημα αν πρέπει κάτι να αλλάξει, σε αυτό έχω απαντήσει ήδη εισηγητικά. Υπάρχει ο κανονισμός του προσωπικού, που κατά τη γνώμη μου είναι ένα πολύ σύγχρονο κείμενο. Και θεωρώ ότι ορθός, καλός και δικαίος για όλα τα θεσμικά όργανα υπάρχει η δυνατότητα εσωτερικών προκηρύξεων, εξωτερικών προκηρύξεων και μετατάξεων. Αν κάποια στιγμή θέλετε φέτος να διοργανώσουμε μια στρογγυλή τράπεζα όπου θα συμμετάσχουν όλα τα θεσμικά όργανα, γιατί ο κανονισμός του προσωπικού ισχύει για όλα τα θεσμικά όργανα, όχι μόνο για την Κομισιόν, τότε βεβαίω εγώ είμαι πρόθυμος, έτοιμος να έρθω εδώ με το επιτελείο μου να επανεξετάσουμε και με τα αντίστοιχα επιτελεία των άλλων θεσμικών οργάνων και να δούμε αν ε, χρειάζονται ο κανονισμός προσωπικού ε, προσθήκες, τροποποιήσεις, βελτιώσεις. Είμαι στη διάθεσή σας για κάτι τέτοιο. Πολύ ευχαρίστως να προσέλθω σε μια τέτοια συζήτηση στρογγυλής τραπέζης. Κύριο Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Κινέζοι λένε ότι πριν κανένας διορθώσει τον κόσμο θα πρέπει να φροντίσει το περιβόλι του, το δικό του το σπίτι δηλαδή. Ή γιατί είχατε για κάποιους διορισμούς ισχυρές αμφιβολίες πριν συμφωνήσατε για την ε, απαλλαγή όσον αφορά τον προπολογισμό του Κοινοβουλίου. Επομένω, όταν κάποιο ε, θέλει κάτι να επικρίνει, θα πρέπει να έχει το απαραίτητο ηθικό κύριο προ τούτο. Έχουμε τώρα τρία ερωτήματα τα οποία προκύπτουν. Πρώτα-πρώτα, έχει τι ε, ικανότητε, ο διοριστής. Δεύτερον, η διαδικασία ήταν διαφορετική από αυτήν που ακολουθήθηκε για τους γενικούς γραμματείς στο παρελθόν και Κατά τρίτον, τηρήθηκαν τα προβλεπόμενα για αυτή τη διαδικασία. κυρία Πρόεδρε, ε, βέβαια έχουν διατυπωθεί διάφορε θεωρίε όσον αφορά την ερμηνεία των κανόνων δικαίου. Και εγώ ξέρω ορισμένε. Υπάρχει η στενή ερμηνεία, υπάρχει η ευρεία ερμηνεία και υπάρχει αυθεντική ερμηνεία. Είναι αυτή στην οποία προβαίνει το Δικαστήριο Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων. Αλλά πάντως το ΔΑΚΙΝΑ, από την Ακρίνη αν η διαδικασία και μας είπε η νομική υπηρεσία ότι υπάρχει αρκετή νομολογία από αυτό σε σχέση με το άρθρο 7 του καταστατικού που αφορά όλα τα θεσμικά όργανα, όσον αφορά δηλαδή τον διορισμό των υψηλών αξιωματούχων. Τρει ερωτήσει, κύριε Πρόεδρε. Πρώτα πρώτα, όσον αφορά τι ικανότητε του Γενικού Γραμματεία. Δεν λέω αν είναι αντιπαθητικό ή συμπαθητικός, εάν έχει φίλους ή εχθρούς, εάν είναι ελκυστικός ή αποθητικός. Ε, κατά πόσο είναι δηλαδή κάποια αξιολογία. Ξέρω ότι υπάρχουν διαδικασίε για ανεξαρτητή αξιολογία, αλλά θα ήθελα να δούμε ακριβώ ε, για ποιο λόγο κατόπιν τη συγκεκριμένη του σταδιοδρομία ε, προήχθη, πώ το λένε, τέλο για αυτή τη θέση. Και μετά, τι έγινε όσον αφορά την, το διορισμό του κυρίου Σελμάγερ, έγιναν τα ίδια ε, σε σχέση με τόσα γίνει στο παρελθόν για του άλλου ΓΓ. Επίση, είχαμε αυτό το ε, ερωτηματολόγιο. Ευχαριστούμε την Κομισιόν για τι απαντήσει έχουμε την ερώτηση παραθμών 133. Λέμε ότι προτίθεται η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στα πλαίσια αυτού του καταστατικού και σε σχέση με τα άλλα θεσμικά όργανα να προβληματιστεί για το πώς μπορεί να προσδώσει περισσότερη διαφάνεια όσον αφορά τους ε, ψήφιους αξιωματούς, όσον αφορά την εξαρτησία, όσον αφορά την ακυρωτητά τους, ε, και γι' τον λόγο να έχουμε περισσότερε δυνατότητε να το ρυθμίσουμε αυτό και τέλο πάντων και περισσότερη ισότητα ευκαιριών στο μέλλον. Κύριε Επίτροπε. Για το ερώτημα για συγκρίσιμους ε, διορισμούς. Από το 2000 είχαμε τρεις διορισμούς γενικών γραμματέων, Σάλιβαν, Ντέι και Όλοι αυτοί οι διορισμοί έγιναν έπειτα από μετάταξη. Από άλλη υψηλόβαθμη θέση, στη θέση του Γενικού Γραμματέα δηλαδή. Ο κύριος Σελμάιερ έχει εξαίρετη ακαδημαϊκή πορεία με επίκεντρο και έμφαση στο Ευρωπαϊκό Δίκαιο. Αλλά Εδώ και 8 χρόνια είναι διευθυντής γραφείου. Ήταν 5 χρόνια νωρίτερα στην ε, τωρινή συνάδελφό σα Βιβιάν Ρέντινγκ και είναι εδώ και 8 χρόνια ε, διευθυντής και συνεργάτης του κυρίου Γιούγκερ. Και πριν από αυτό ήταν, όπως είπα, στο επιτελείο της κυρίας Ρέντινγκ συμμετέχει και εργάζεται εδώ και πάνω από 10 χρόνια λοιπόν στην Κομισιόν. Και θέλω να τονίσω για άλλη μια φορά. Διευθυντής επικεφαλής του γραφείου Επιτρόπου είναι ίση θέση με τη θέση του Διευθυντού και επικεφαλής γραφείου του Προέδρου της Κομισιόν είναι ισάξια η θέση αυτή με τη θέση ενός Γενικού Διευθυντή. Από αυτή την άποψη λοιπόν επρόκειτο για μετάταξη στο ίδιο επίπεδο και στο ίδιο μισθολογικό επίπεδο. Δεν βγάζει περισσότερα χρήματα αυτή τη στιγμή ο κύριος Σελμάιρ σε σύγκριση με αυτά που έβγαζε πριν από το διορισμό του στη θέση του Γενικού Γραμματέα. Ja, danke, Frau Vorsitzende. Κύριος Κούν, ευχαριστώ Κύριε Επίτροπε, σα ευχαριστώ για τις ε, απαντήσεις σας και για την προσφορά που μας κάνατε να προσέλθετε σε μια συζήτηση στρογγυλή τραπέζη. Νομίζω ότι είναι αναγκαίο κάτι τέτοιο. Όλοι από κοινού, όλα τα θεσμικά όργανα να εξετάσουν πώς θα, θα μπορούσαμε να αποφύγουμε τέτοια φαινόμενα στο μέλλον. Σε σχέση με το άρθρο 7 ε, θεωρώ ότι ε, είναι ένα άρθρο το οποίο οπωσδήποτε πρέπει να τροποποιηθεί και να ασαφινιστεί προκειμένου να ε, ορίζεται συγκεκριμένα ο αριθμός των υποψηφίων που πρέπει να υπάρχει, η διαδικασία που πρέπει να ακολουθείται, ο χρόνος που θα πρέπει να αφιερώνεται στη διαβούλευση και στη συζήτηση και να μην μπορεί να γίνουν τέτοιες προαγωγές μέσα σε λίγα λεπτά. Και επαναλαμβάνω αυτό που είπε και η συνάδελφος ε, από την νομική υπηρεσία ότι βάσει του άρθρου 4 πρέπει να υπάρχει εξωτερική προκήρυξη της θέσης εκτός αν υπάρχουν συγκεκριμένες περιστάσεις οι οποίες να δικαιολογούν το αντίθετο. Εγώ ε, βεβαίως νομικός, ε, με τη νομική ασχαλούμε ε, και μόνο. Ε, ήταν πολύ εντυπωσιακά όμως αυτά που μας είπατε. Να μας πείτε σας παρακαλώ ποιε ακριβώς ήταν αυτές οι εξαιρετικές περιστάσει, γραπτό παρακαλώ σε απάντησή σας, ποιε ήταν αυτές οι εξαιρετικές περιστάσει που σας οδήγησαν να λάβετε αυτήν την κατεξαίρεση απόφαση σε σχέση με το διορισμό του συγκεκριμένου ανθρώπου στη θέση του Γενικού Γραμματέα. Επίτροπο. Θα μπορούσαμε να συμφωνήσουμε ποια ακριβώς, να μας ενημερώσετε κι εσείς ποια ακριβώς είναι τα θέματα, ε, ποια είναι τα άρθρα του κανονισμού προσωπικού που θα θέλατε να τροποποιηθούν και να το συζητήσουμε. Ως προς την μετάταξη και τις πληροφορίες που ζητάτε, δεσμεύομαι ότι εντός 10 ημερών θα σας απαντήσω. Για τον χρόνο συζήτησης και διαβούλευση Η απάντηση μου είναι και ναι και όχι. Στην ελεύθερη αγορά για παράδειγμα μπορεί κανείς να μάθει ότι η Deutsche Bank αναζητά νέο διευθυντή. Αν μάλλον υπήρχε μια τέτοια δυνατότητα, θα βλέπατε την ε, μετοχή της Deutsche Bank να καταραίει. Όταν λοιπόν ο κύριος ε, Juncker μου είπε εμένα και στον κύριο Τίμερμανς ότι ο Ιταλιάνερ φεύγει, θεωρώ ότι πρέπει να τον αντικαταστήσει ο Σελμαϊρ. πιστεύετε ότι σε περίπτωση που σε αυτή τη φάση εμείς αρχίζαμε μια δημόσια συζήτηση αυτό θα ωφελούσε την Κομισιόν και την Ευρωπαϊκή Ένωση συνολικά ή όχι. Νομίζω όχι. Δεν βοηθάει μια τέτοια διαδικασία. Και αντίστοιχε διαδικασίε βεβαίω ε, ακολουθούνται και σε όλου του διεθνεί οργανισμού και στι ε, πολιτικέ ομάδε. Πρόεδρο, για ποιο λόγο σύμφωνα με το άρθρο 7 δεν πήρε μαζί του τη θέση όμως αυτό είναι το, ερώτημα. Ο κύριος Λούκε έχει το λόγο. Ευχαριστώ. Τρεις ερωτήσεις θέλω να θέσω. Πρώτον, το άρθρο 10 του καταστατικού ορίζει ότι κάθε ε, υπάλληλο πρέπει να ε, ε, ενεργεί με τρόπο που θα ε, προστατεύει την ακαιρεότητά του. Ο κύριος Σέλμαερ όμως έχει μιλήσει για ε, μαλάκες, για δημοσιογράφους με αυτόν τον τρόπο. Το ερώτημα μου, κύριε Επίτροπε, αυτά, αυτές τις δηλώσεις του κυρίου Σέλμαερ τις ελέγξατε ως Επιτροπή. Το σώμα των Επιτρόπων ενημερώθηκε για αυτές τις ενέργειες του κυρίου Σέλμαερ και τις δηλώσεις του σε δημοσιογράφο. Φαντάζομαι ότι δεν είχατε λάβει γνώση ε, αυτήν, ε, αυτών των ε, γεγονότων. Γιατί κάτι τέτοιο είναι ασύμβατο με το άρθρο 12. Δεύτερο ερώτημα. Το άρθρο 17 ορίζει ότι ο υπάλληλο δεν επιτρέπεται να κοινοποιεί πληροφορίε των οποίων λαμβάνει γλώσση στο πλαίσιο της εκτέλεσης των καθηκόντων του. Ωστόσο, ο ε, δημοσιογράφος Μούλερ του Σπίγκελ ισχυρίζεται ότι ο κύριος Σελμαέρ πολλές φορές του έχει διαβιβάσει και κοινωνιποιήσει τέτοιες εμπιστευτικές πληροφορίες. Το Σώμα των Επιτρόπων έλαβε γνώση, ενημερώθηκε σχετικά με την παραβίαση του κανόνα αυτού του άρθρου 17 από τον κύριο Σέλμαϊ. Επίσης, σύμφωνα ε, με ιδεσιογραφικά δημοσιεύματα ο ίδιος ο κύριος Σελμάιερ φέρεται να ε, εξοράισε το άρθρο της Wikipedia στις 29 Δεκεμβρίου του 2017. Ο ίδιος. Το ερώτημά μου είναι πότε το Σώμα των Επιτρόπων έλαβε τα έγγραφα, τα δικαιολογητικά έγγραφα για την, ε, για την υποψηφιότητα του κυρίου Σελμάιερ. Είχατε χρόνο να επαληθεύσετε τις πληροφορίες που περιλαμβάνονται σε αυτές. Μπορέσατε να ε ε, ε, ε, βεβαιωθείτε ότι ε, ο κύριος Σελμάιερ δεν αξιοποίησε τη Wikipedia προκειμένου να εξοραίσει τη δική του θέση και το πρόσωπό του ενώπιον του Σώματος των Επιτρόπων, το οποίο θα συζητούσε για τον ίδιο, κύριε Λούκερ. Λούκε. Αν πράγματι ο κύριος Μούλερ αποκλήθηκε με αυτή τη λέξη από τον κύριο Σέλμαερ, προφανώς δεν πρόκειται για κάτι κομψό ή κάτι σωστό. Εμείς ως Κομισιόν δεν ρωτήσαμε τον κύριο Μίλλερ αν πράγματι διεμήφθησαν τα πράγματα με αυτόν τον τρόπο, ούτε βεβαίω ε, συζητήσαμε για αυτό το θέμα κατά τη συζήτηση της υποψηφιότητα του κυρίου Σέλμαερ. Βεβαίω, καθένα πρέπει να ελέγχει και αυτά που λέει και τον τρόπο με τον οποίο ενεργεί και πράττει στη δημοσιότητα. Προκειμένου να μην ε, προσβάλλεται ε, να μην προσβάλλονται τρίτοι. Θεωρώ όμως ότι κάθε υποψήφιος έχει το δικαίωμα να ε, εξετάζεται για τη συνολική του παρουσία. Ο κύριο Σελμαΐρ βεβαίω έχει αδύναμα και δυνατά σημεία. Θεωρώ όμω ότι τα δυνατά σημεία του υπερέχουν των αδύναμων σημείων του και νομίζω ότι υπό το φως των ε, εξαιρετικών του ικανοτήτων μπορούμε να του αναγνωρίσουμε ότι έχει ως άνθρωπος δικαίωμα να έχει και κάποιες αδυναμίες. Εγώ λοιπόν δεν θεωρώ ότι έχει ε, παραβιάσει ποτέ την υποχρέωση εμπιστευτικότητας που τον δεσμεύει. Η Wikipedia δεν είναι το μητρό προσωπικού της Κομισιόν. Οποιοςδήποτε μπορεί να μπει στην ε, Wikipedia και να προσθέσει στοιχεία σε σχέση με το βιογραφικό του ή και να τα αλλάξει. Και με την ευκαιρία Αφού διάβασα σχετικά δημοσιεύματα, εγώ διαπίστωσα τις αλλαγές που είχαν γίνει στη Wikipedia. Οι δικές μας εξελ, ε, αξιολογήσεις προσωπικού εδράζονται σε, στις εκθέσεις που λαμβάνουμε από τους εκάστοτε προεσταμένου των εργαζομένων, των υπαλλήλων. Αυτές οι εκθέσεις αξιολόγησης αρχιοθετούνται και στη συνέχεια χρησιμοποιούνται και αξιοποιούνται στις διαδικασίες επιλογής προσωπικού. Στον κύριο Σέλμαϊερ υπήρχε ε, προκήρυξη για τη θέση του αναπληρωτή γενικού γραμματέα. Ενημερωθήκατε κι εσείς γι' αυτό. Είχαμε λάβει την υποψηφιότητά του, τα δικαιολογητικά του. Αυτά υπάρχουν στη Γενική Διεύθυνση Ανθρώπινου Δυναμικού, τη δική μου Γενική Διεύθυνση, αλλά δεν διαβάζονται άμεσα σε όλο το σώμα των, επιτρέ... επιτρόπων, αλλά ξεκινά μια διαδικασία με assessment center και εσωτερική διαδικασία, η οποία και ακολουθήθηκε. Και σας είπα ότι σε ε, ασφαλή αίθουσα εκπρόσωποι της Επιτροπής σας μπορούν να έχουν πρόσβαση σε αυτά τα έγγραφα και αφού ολοκληρωθεί αυτή η διαδικασία υποβάλλεται πρόταση στο Σώμα των Επιτρόπων. Αυτή είναι και η διαδικασία που ακολουθήθηκε, αυτή τη φορά. κύριος Λούκε, δεν απαντήσατε πότε λάβαν οι επίτροποι τα δικαιολογητικά του κύριου Σέλμαϊρ. Απαντήστε παρακαλώ. Και δεύτερον, δεν είναι υποχρέωσή σας να ελέγχετε αν ε, κάποιος υπάλληλο έχει παραβιάσει το καταστατικό και τον κανονισμό προσωπικού. Το δεύτερο το ελέγχουμε αν υπάρξουν στοιχεία που να τεκμηρώνουν κάτι τέτοιο ή αν έχουν υπάρξει σχετικές ενδείξεις ή και καταγγελίες παράπονα, τότε θα λάβουμε τα αναγκαία μέτρα. Αλλά εξ όσων γνωρίζω δεν έχει συμβεί κάτι τέτοιο. Τα έγγραφα του προσωπικού, τα δικαιολογητικά των υποψηφιότητων βρίσκονται πάντοτε στη διάθεση των ε, εξεταστικών επιτροπών το Σώμα των Επιτρόπων όμω ενημερώνεται στη συνέχεια από εμένα προσωπικά, προφορικά και λαμβάνει μια σύνοψη των πληροφοριών αυτών. Αυτό ακριβώς έγινε και την Τετάρτη 21 Φεβρουαρίου. Κύριε Τρεμόζα. Δεν έχει ανάψει το μικρόφωνο ο κύριος Τρεμόζα. Μικρό. Δεν λειτουργεί το μικρόφωνο του Τρέμος. Entschuldigung. Συγγνώμη, συγγνώμη, κύριε Τρεμόζα. Κύριε Επίτροπε, σας καλωσορίζω για άλλη μια φορά εδώ στο Κοινοβούλιο. Ως Επίτροπος, κάνατε πολύ καλή δουλειά. Ε, θυμάμαι ότι το 2013 είχα ζητήσει συνάντηση μαζί σας, με σας και με το επιτελείο σας. Και το ερώτημά μου είναι, πού είναι ο κύριος Γιούγκερ, γιατί δεν είναι εδώ να απαντήσει στις ε, ερωτήσεις μας ο κύριος Γιούγκερ. Γιατί συνδέεται το όνομά σας με το Selmayr Γκέιτ; Έχω τις εξής ερωτήσεις. Πώς ήταν τον ο καλύτερος των υποψηφίων ο κ. Σελμαγιάννη είναι ο μόνος υποψήφιος. Πώς θα εξηγήσουμε στους Ευρωπαίους ότι έχουμε μόνο έναν υποψήφιο. Πού πήγε η αξιοπιστία. Πώς τα, πώς τα παιδιά μου. Μελετήστε. Σκληρά. Γιατί από το αν θα μελετήσετε τώρα θα το αν θα έχετε μια πολύ καλή δουλειά αύριο. Επομένως αυτό για μαυρώσει την ε, φήμη της Ευρωπαϊκής Άλλη ερώτηση συμμετέσχε στην αξιολόγηση των ε, απαντήσεων που δώσατε στο Κοινοβούλιο. Θέλω μια απάντηση ναι ή όχι. Διότι εάν συμμετέσχε στην απάντηση του ερωτηματολογίου, αυτό αποτελεί παραβίαση του άρθρου 11. Άρα απαντήστε μου ναι ή όχι. Συμμετέσχε ή όχι στις απαντήσεις. Επίσης, και κάτι άλλο θέλω να σας πω, γιατί η Νέσα Γιάλα σας ρώτησε για την συμμετοχή του σε μια συνάντηση του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος και είπατε ότι δεν έχετε ιδέα. Πρόκειται για την 23η Μαρτίου. Αλλά σε άλλη απάντηση είπατε ότι ήταν εκεί εκτός αίθουσας ε, δεν καταλαβαίνω. Πέστε μας, μπήκε ή όχι στην αίθουσα σε εκείνη την συνάντηση του ΕΛΚ. Ο Επίτροπος Ακριβώς επειδή για να απαντήσουμε στα ερωτήματά σας χρειάστηκαν οι πληροφορίες ε, του κυρίου Σελμάιερ, βεβαίως συμμετείχε στις συζητήσεις που έγιναν για τη σύνταξη των απαντήσεων και προσωπικά. Αυτό όμως δεν το έκανε προκειμένου να επηρεάσει τις διατυπώσεις, αλλά για να συμπληρώσει και να καταστούν όσο το δυνατόν πιο ολοκληρωμένες οι απαντήσεις. Wenn eine Frage gewesen war, ab wann wusste Martin Μα όταν θέτεται ερώτημα, πότε το ήξερε αυτό ο κύριος Σελμάιρ, από πότε είχε λάβει γνώση αυτό, του στοιχείου. Αν ήταν 15, 2016, 2017, Ιανουάριος, Φεβρουάριος, Μάρτιος, μα προφανώς ποιος άλλος μπορεί να απαντήσει αυτό το ερώτημα, αν όχι ο ίδιος ο κύριος Σελμάιερ. Αν απαντούσαμε, μα συγχωρείτε δεν ξέρουμε, έχουμε βεβαίω τον Γενικό Γραμματέα εδώ, που είναι στον πάνω όροφο, αλλά δεν μπορούμε να σας απαντήσουμε στο ερώτημά σας ε τότε θα ήθελα να δω πώς θα είχατε αντιδράσει. Γιατί τώρα γελάτε. Τότε όμως θα έπρεπε να μας, να μας, να μας γελιοποιείτε. Αν είχαμε κάνει κάτι τέτοιο. Γι' αυτόν τον λόγο συζητήσαμε με τον ίδιο τον κύριο Σελμαϊρ, λάβαμε τις πληροφορίες αυτές από τον ίδιο τον κύριο τον Σελμαϊρ, ακριβώς για να μπορέσουμε να σας δώσουμε όσο πιο ολοκληρωμένη απάντηση μπορούσαμε. Δεν είπα ποτέ ότι είναι ο καλύτερος. Είπα ότι έχει υψηλές ικανότητες, υψηλά προσόντα και ότι είναι κατάλληλος υποψήφιος για τη θέση στην οποία διορίστηκε. Τρίτον, είπατε που είναι ο κύριος Γιούγκερ. Εγώ ε, γνωρίζω ότι ε, έχει ανηλυμένες υποχρεώσεις. Ήταν μέχρι χθε στη Βάρνα, γύρισε σήμερα στις, 3 ε, το, γύρισε το πρωί και όταν λάβαμε την επιστολή από την Επιτροπή σας, αυτή απευθυνόταν στον κύριο Έτιγκερ, ούτε στον κύριο Σελμάιρ, ούτε στον κύριο Γιούνκερ. Κάτι αντίστοιχο έγινε και στο Στρασβούργο. Η διάσκεψη των Προέδρων προσκάλεσε εμένα προσωπικά. Και εγώ στο κοινοβούλιο έρχομαι όποτε μου απευθύνεται πρόσκληση. Αν δεν μου έχετε απευθύνει πρόσκληση, δεν έρχομαι. Εγώ δεν είπα no idea, ότι δεν έχω ιδέα. Απάντησα στο ερώτημα της Αγιάλα Σέντερ ότι υπήρξε κομματική συνάντηση. Είπα ότι δεν μπορώ να απαντήσω. Ακριβώς γιατί γίνονται χιλιάδες τέτοιες κομματικές ε, συνεδριάσεις πριν από τις ή ή και στο περιθώριο των συνόδων κορυφής. Όταν όμως διευκρίνησε ότι επρόκειτο ότι μίλησε, ότι μιλούσε για την συνάντηση του ΕΛΚ την προηγούμενη εβδομάδα, απάντησα ότι βρισκόταν μαζί με το επιτελείο του στο κτίριο του Συμβουλίου, αλλά όχι στην ίδια αίθουσα που βρίσκονταν οι πρόεδροι του ΕΛΚ. Ήταν έξω από την αίθουσα, μπροστά από την πόρτα, ακριβώς διότι ήταν απαραίτητο να μπορέσει να παράσχει τις συμβουλές του βάσει και των εξελίξεων που θα είχαμε εκείνη τη μέρα και εκείνες τις ώρες σχετικά με την υποβολή δασμολογικών μέτρων από πλευράς ΕΠΑ. Ήταν μαζί με τον επικεφαλής του γραφείου της κυρίας Μέρκελ, του γραφείου του κυρίου Τούσκ και με όλους τους υπόλοιπους ε, διευθυντές γραφείων. Άλλες τρεις ομιλητές έχουμε, κύριο Σάβαμα. Thank Σας ευχαριστώ, Πρόεδρε. Αυτή θα είναι η τελευταία μου παρέμβαση σε αυτή τη συνεδρίαση. Επομένως, θα ήθελα εσκεμένα να επαναλάβω τα όσα είπα στην αρχική μου παρέμβαση και στις αρχικές μου παρατηρήσεις. Υπάρχει μια σαφής τάση, εσκεμένη θεωρώ, να προσπαθείτε να μας πείτε ότι η ακαιρεότητα και η διαφάνεια είναι το ίδιο πράγμα. Σε καμία περίπτωση. Όπως σας είπα, αλληλοεπικαλύπτονται σε πολλές περιπτώσεις. Και στη συγκεκριμένη περίπτωση συμβαίνει κάτι τέτοιο. Ωστόσο, και θα ήθελα εδώ πέρα να αναφερθώ σε κάποια από αυτά που ακούσαμε σήμερα, και αυτό έχει να κάνει πραγματικά με τη διαφορά την ειδοποιώ ανάμεσα στην ακαιρεότητα και τη διαφάνεια. Αναφέρομαι σε εσά κύριε Γκερμπράντι. Δώστε την εντύπωση ότι εμπλέκεται ο κύριος Γιούνκερ σε μία παράνομη συνωμοσία, σε ένα Watergate 2, όπου βρέθηκε τότε κάποιος υπεύθυνος να έχει παρανομήσει τελικά, να έχει παραδεί τον νόμο ενώ στη συγκεκριμένη περίπτωση δεν μπορεί να υποθεί κάτι τέτοιο, τουλάχιστον μέχρι στιγμή. Θα δούμε. Θα δούμε πώ θα εξελιχθούν τα πράγματα. Κύριε Στάε, είπατε κι εσεί, απευθυνόμενο προ τον Επίτροπο Έντιγκερ, Μπάρτ, συγγνώμη, πρέπει πραγματικά να αναφέρω αυτό το οποίο είπε. Είπατε στον Επίτροπο Έντιγκερ ότι δεν συνειδητοποιείται την ζημία που έχει γίνει για την φήμη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής όταν η λεγόμενη αυτή καζόμενη ζημία ουσιαστικά έχει να κάνει μόνο με τις ε, πολύ επιθετικές ε, καταγγελίες που έχουν γίνει κυρίως από τους ίδιους τους πρασίνους. Πρόκειται για μία παγιωμένη τακτική που έχετε προκειμένου να παρουσιάσετε τα πράγματα με το δικό σας τρόπο. Ουσιαστικά εδώ πέρα έχουμε μια αυτοεκπληρούμενη προφητεία η οποία δεν έχει καμία ε, θέση θα έλεγα στη συζήτηση που κάνει η Επιτροπή αυτή και ιδίω στι περιπτώσει εκείνε που αλληλοπικαλύπτονται ακαιρεότητα και διαφάνεια. Ο κύριος Βον είπε ουσιαστικά αυτό το οποίο λέω και εγώ. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα πρέπει να στείλει ένα μήνυμα αυτή τη στιγμή ότι κατανοεί την κριτική που τη γίνεται και ουσιαστικά έχει να κάνει αυτό με τη διαφάνεια και με την τροποποίηση των κανόνων για το μέλλον. Ακριβώς επειδή στο σημερινό κόσμο δεν μπορούμε να ανεχτούμε τέτοιες πρακτικές. Δεν έγινε κανένα έγκλημα όμως και κάτι ολοκληρώνοντας την παρέμβασή μου και τον έφερε και ένας συνάδελφος, ο κύριος Βόνα, δεν κάνω λάθος πριν από λίγο. Πραγματικά είναι λυπηρό, λυπηρό ότι έχουμε μόνο τον Επίτροπο Έτιγκερ εδώ μαζί μας αρχίζω και λυπάμαι για αυτά που είπα στους συντονιστές. Εγώ τον ε, κύριο Γιούγκερ ενδεχομένω θα ήθελα να έχω εδώ πέρα ή τον κύριο Σέλμαερ τον ίδιο και όταν μην ταλαιπωρούμε τον κύριο Έτιγκερ γιατί ε, ουσιαστικά έπρεπε να αντιμετωπίσει μια συγκεκριμένη απόφαση, ένα γεγονό το οποίο ελήφθη υπόψη μία μέρα πριν τη συνεδρίαση των, του σώματο των Επιτρόπων. Ο Επίτροπος έχει το λόγο. Κυρία Πρόεδρε, κύριοι Ευρωβουλευτέ, σημειώνω ότι το ερώτημα σχετικά με τη διαδικασία θα απαντηθεί γραπτώς εντός των επόμενων δέκα ημερών. Θα σας αποστείλουμε γραπτή απάντηση στην Επιτροπή σα. Α, συγγνώμη, έχετε και άλλε ερωτήσει Γιατί ε, πιέζομαι χρονικά. Ο κύριο Πανιού. Ε, κύριε Επίτροπε, κυρία Πρόεδρε, συνάδελφοι, πάνω από δύο ώρε βρισκόμαστε εδώ στη συνεδρία τη Επιτροπή Ελέγχου του και έχουμε αυτόν τον αγώνα πινκ-πονγκ να μας απαντάει ο κύριος Έτιγκερ συνεχώς θα μπορούσατε να κάνετε καριέρα στο σινεμά, κυρία Τιγκέρ. Μόλις θα φύγετε από το Σώμα των Επιτρόπων. Και είναι μεγάλη ταλαιπωρία εδώ και δύο ώρες τον ακούμε όλα αυτά τα οποία ακούμε. Όχι, όχι, όχι, ποτέ δεν συμμετέσχε στην επίμαχη συνεδρία ο κύριο Ζελμαγέρ. Μετά λέτε. Μα όχι, όχι. Αυτό, αυτό. Ε, δεν μπορούσε να αφήσει το πλευρό του Πρόεδρου της Κομισιόν. Ε, θυμάστε τον ε, Μαζαρίνα, τον Καρδινέλιο που ήταν επί μια εικοσαετία πρωθυπουργός επί Λουδοβίκου 14 στη Γαλλία. Δεν ναι. νομίζω ότι ο κύριος ε, Γιούνκερ είχε το ίδιο πρόβλημα όπως είχε τότε τόσα χρόνια ο Λουδοβίκος ο 14ος. Μα τέτοια ε, ε, εντύπωση μας δίνει το ότι ε, αυτός ο σούπερ σύμβουλος ήταν απαραίτητος τόσα χρόνια δίπλα στον Γιούγκερ και άρα θα έπρεπε να βρίσκεται στην πρώτη γραμμή αδιαφορώντας για κάθε πρωτόκολλο, κάθε κανόνα. Μα έχουμε και τη γνωμοδότηση της νομικής υπηρεσίας που ξεκαθαρίζει το ότι υπάρχει νομικό πρόβλημα σε αυτόν τον διορισμό ως γάμα γάμα του κ. Σελμαγιάς. Και μας είπε για την πάγια νομολογία η νομική υπηρεσία. Δεν έχουμε ιδιαίτερο πρόβλημα σύγκρουση συμφερόντων κλπ. κλπ. Μα τι, λάθος κάνει, δεν λειτουργεί εύρεθμα η νομική υπηρεσία. δεν και εσείς κύριε Πρόεδρε. Εδώ έχουμε δύο βασικά ζητήματα. Βρισκόμαστε στα πρόθυρα των ευρωεκλογών και παντού, παντού βλέπουμε ε, το πόσο ανεβαίνει η επιρροή των εθνικιστών, των αντιευρωπαίων. Ε, τι θα πει ο κόσμος για το αν ωφελεί, αν, αν είναι χρήσιμη η Ευρωπαϊκή Ένωση. Γιατί να υπάρχει Ευρωπαϊκή Ένωση με όλα αυτά τα οποία κάνετε. Άρα δεν να αμφιβόλο η Ευρωπαϊκή Οικοδόμηση είναι νομικό θέμα αλλά και πολιτικό θέμα. Σημαντικό. Μα αυτό είναι πολιτική τύφλωση κύριε Επίτροπε να μην μπορείτε να δείτε το πόσο σημαντικές είναι οι πολιτικές συνέπειες. Πάνω σε αυτό απαντήστε μας όσον αφορά τον διορισμό στις πολιτικές συνέπειες αυτής της ε, παράτυπης, παράνομης τέλος πάντων ε, του διορισμού αυτού. Εμάς είμαστε υπεύθυνοι οικοδόμηση. Θα πρότεινα να δώσουμε το λόγο και στον συνάδελφο Στεχόφσκι. Ε, Ευχαριστώ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Κύριε Πίτροπε, δεν θα ήθελα να επαναλάβω τα όσα υπόθηκαν. Ήδη πολλές ερωτήσεις έχουν απαντηθεί. Θα είμαι πολύ σύντομος. Και θα ήθελα να μου δώσετε μια απάντηση στην ακόλουθη ερώτηση, κύριε Πίτροπε. Ποιο δίδαγμα έχετε αντλήσει από την όλη συζήτησή μας. Υπάρχει κάτι που έχετε μάθει σήμερα, το οποίο θα μπορέσει να εφαρμόσετε αν μη τι άλλο στο μέλλον. Θα ακολουθήσετε και στο μέλλον τις ίδιες διαδικασίες Πιστεύετε πραγματικά ότι ήταν ορθές οι διαδικασίες οι οποίες ακολουθήθηκαν και ποια είναι η προσωπική σας τώρα άποψη βλέποντας την ε, κα, κατακραυγή αυτή που υπήρχε εναντίον, τη της απόφασης αυτής, την κατακραυγή δηλαδή από την κοινή γνώμη. Πιστεύετε πραγματικά ότι η διαδικασία που μας παρουσιάσετε εδώ πέρα σήμερα ήταν όντως διαφανή. Σας ευχαριστώ. Επίτροπος. Δεν θέλω να κάνω ανακοινώσει για το τι προτιθέμεθα θα να κάνουμε στο μέλλον, αλλά πρέπει να σας πω, ηθοποιός δεν είμαι. Νομίζω ότι ήταν αρκετά δραματική η παρέμβασή σας. Όταν λέτε ότι υπάρχουν νομικά κενά, σας ευχαριστώ την προσοχή. Τηρήσαμε τον κανονισμό του προσωπικού που κι εσείς έχετε συναποφασίσει και θεσπίσει. Υπάρχει, υπάρχουν μόνο δύο απαντήσεις. Ναι και όχι. Συμφωνούμε ότι ακολουθήθηκαν όλες οι διατάξεις του κανονισμού προσωπικού. Κάποιοι είπαν ότι ακολουθήσαμε το γράμμα αλλά όχι το πνεύμα ή το πνεύμα εν μέρη μόνο. Εγώ διαφωνώ. Αλλά και πάλι δεν έχουμε παραβίαση των κανόνων. Καταλαβαίνω ότι υπάρχει μια δυνατότητα ερμηνείας από το Κοινοβούλιο. Και μάλιστα υπάρχει και η δυνατότητα να υπάρχουν και πολλές ερμηνείες. Όμως το ερώτημα είναι σαφές. Ο κανονισμός προσωπικού τηρήθηκε, τηρήθηκε. Κατά γράμμα, κατά γράμμα. Γι' αυτό και επαναφέρω την πρότασή μου. Να προχωρήσουμε σε μια συζήτηση της Ογγλής Τράπεζας, στην οποία θα συμμετέχουν όλα τα θεσμικά όργανα και να εξετάσουμε πιθανές βελτιώσεις στον κανονισμό του προσωπικού. Πάντως, σήμερα νομίζω ότι κανείς προφανώς δεν μπορεί να είναι ιδιαίτερα ευτυχής με τα όσα συνέβησαν τις προηγούμενες εβδομάδες. Ας εξετάσει όμως καθένας αυτοκριτικά κατά πόσο συνέβαλε στην ουσιαστική συζήτηση, στην αντικειμενικότητα με την οποία διεξήχθη η συζήτηση. Τα ερωτήματα που πρέπει να μας απασχολήσουν είναι δύο. Έχει τα τυπικά και προσωπικά προσόντα ο κύριος Σέλμαϊρ για να καλύψει τη θέση στην οποία διορίστηκε. Και δεύτερον, η Κομισιόν ακολούθησε τους προβλεπόμενους κανόνες. Εγώ λέω χωρίς καμία επιφύλαξη και στα δύο ερωτήματα ναι. Αλλά βεβαίως μπορείτε κι εσείς να κρίνετε την απάντησή μου αυτή και να δώσετε τη δική σας απάντηση. Επαναλαμβάνω ότι μέσα στις επόμενες δέκα μέρες θα σας αποστείλουμε γραπτός την απάντησή μας σχετικά με τις, ε, ε, με τα βήματα που ακολουθήθηκαν. Θα επιμείνω να γίνει αυτή η συζήτηση της Ρογγυλής Τραπέζης πριν από το καλοκαίρι και επαναφέρω και την πρότασή μου σε αίθουσα στα κτίρια της Κομισιόν να παρέχουμε πρόσβαση στα μέλη της Επιστροπής σας στα δικαιολογητικά της υποψηφιότητας του κυρίου Σέλμαϊρ κύριος Τάραντ. Ποτέ δεν είδα να είναι τόσο δυναμικός, τόσο ορμητικός ο καλός βίος του κύριος Σαρβάμα. Δεν ξέρω. Άρχισε να αμφιβάλλω. Δεν ξέρω αν θα ρίξω λάδι στη φωτιά ή αν αυτό θα να είναι πιο πολύ κατευναστικό. Και θέλω κάτι να ρωτήσω. Όχι τον κύριο Έτιγκερ γιατί έχει καθήκον να υπερασπιστεί αυτή την απόφαση, είναι ένας μεγάλος ωραίος μαχητής και επειδή όλες αυτό κάνει. Και στις 3 η ώρα ήμασταν 175 εδώ μέσα και δεν μετράω τους διερμηνείς και συζητούσαμε για τον διαβόητο Σέλμαγερ. Είναι αυτό αποτελεσματικό, δεν ξέρω. Τέλος πάντων, η παρατήρηση που εγώ βγάζω από όλα αυτά είναι η εξής. ερώτημα προς όλους εμάς τι μπορούμε να κάνουμε ούτω ώστε να αποφύγουμε το να ξανασυμβούν τέτοια πράγματα. Βέβαια δεν έχω τη χαρά την τιμή να γνωρίζω προσωπικά τον Δεσσερ Μάγερ, αλλά από τον Φρεντρίκο το Μεγάλο μάλλον ε, δανείστηκε το ότι όταν κανείς έχει την δυνατότητα να κατακτήσει κάτι πρέπει να το κάνει ευθύ αμέσω. γιατί οι νομικοί και οι ιστορικοί θα σε δικαιώσουν. Όμως για μας είναι αυτό η πιο σωστή στρατηγική. Μα αν ο ίδιος ετοίμασε τις απαντήσεις του ερωτηματολόγιο, ε, α έρθει να βοηθήσει από κοντά. Τέλος πάντων. Ωραία, ωραία η συζήτηση που κάναμε. Και ας βεβαιωθούμε ότι είμαστε σωστοί σε αυτή τη συζήτηση, γιατί υπάρχουν σύννεφα που μαζεύονται στον ορίζοντα. Πάμε τι, για εμπάργκο όσον αφορά τον ορισμό του Πρόεδρου της Ευρωπαϊκής και των Επιτρόπων. Αν υπάρχει τέτοιου είδους σύνεβο θα πρέπει να το ξεκαθαρίσουμε και να κάτσουμε να τα διαπραγματευτούμε πριν αυτά όλα κρυθούν. Εδώ. Καλά, άντε, άντε, να βάλω τελεία εδώ. Πρόεδρος. Ευχαριστώ. Και ολοκληρώσαμε το θέμα αυτό. Για το επόμενο θέμα πρέπει δυστυχώς να σας πω ότι το σχέδιο ψηφίσματος δεν έχει ε, καταρτιστεί ακόμα, δεν έχει συνταχθεί ακόμα. Ε, θέλουμε να συμπεριλάβουμε στο ψήφισμα αυτό και τις, ε, τα συμπεράσματα της σημερινή μας συζήτησης. Διάφορα υπάρχουν, όχι. Α, Μπάρτ, παρακαλώ. Να απαντήσω σε αυτό που είπε ο κύριος Σάβαμα. σχετικά με τη στρατηγική των πρασίνων. Κύριε Σάβαμα, θα σας συμβούλευα να ξαναδείτε τη συζήτηση που έγινε στην Ολομέλεια και να ακούσετε τι είπε η κυρία Γκροστέτ, τι είπε ο κύριος Βέρνερ Λάγκερ από τους Γερμανούς ε, Χριστιανοδημοκράτες για τον κύριο Σέλμαερ και μετά να εξετάσετε τη δική σας στάση. Θα δείτε λοιπόν ότι δεν είναι μόνο οι πράσινοι αυτοί που εξέφρασαν τις αμφιβολίες τους και τις ανησυχίες τους για τη διαδικασία. Eh, Ευχαριστώ Πρόεδρε. Κάτι για την πολιτική μου ομάδα. Θα ήθελα να στηρίξω τα όσα είπε μόλις τώρα ο κύριο Στάε. Υπάρχει μια γενικότερη ανησυχία και υπάρχει και κάτι διαδικαστικό. Σαφώς μπορούμε να συζητήσουμε την πρόταση ψηφίσματος όταν τη λάβουμε. Αλλά υπάρχουν ακόμα πολλά ερωτήματα τα οποία εκκρεμούν, κύριε Πρόεδρε. Δεν αφέρθηκε, για παράδειγμα, ο Επίτροπος στο άρθρο στην εφημερίδα Λεσουάγα όπου α, εκεί πέρα ο κύριο Σελμάιρ παραδέχθηκε ότι του είχε προσφερθεί το πόστο αυτό από τον κύριο Γιούγκερ πριν τα Χριστούγεννα. Υπάρχει το ζήτημα αυτό, αλλά υπάρχουν και άλλα κρεμή ερωτήματα τα οποία δεν απαντήθηκαν από τον Επίτροπο. Νομίζω λοιπόν ότι πολύ γρήγορα θα πρέπει να συντάξουμε ένα νέο ερωτηματολόγιο το οποίο θα πρέπει να απευθύνουμε στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ωραία. Να βάλουμε λοιπόν μια προθεσμία για την υποβολή των νέων ερωτημάτων. Ας προσπαθήσουμε λοιπόν μέχρι το Πάσχα να αποστείλουμε τον νέο μας κατάλογο με, προς την Κομισιόν προκειμένου να προετοιμαστούμε και για τροπολογίες ενόψει της Ολομέλειας. Συγγνώμη και λυπάμαι που το ψήφισμα δεν είναι έτοιμο ακόμη, αλλά είναι σημαντικό να εξασφαλίσουμε ότι θα είναι και ουσιώδες αυτό το ψήφισμα. Γι' αυτό και χρειάστηκε να συμπεριλάβουμε διάφορες πληροφορίες, διάφορα στοιχεία, να συμπεριλάβουμε, αποφασίσαμε και, τις, ε, και τα συμπεράσματα της σημερινής συζήτηση με τον Επίτροπο και από εκεί και πέρα ε, θα προχωρήσουμε στη σύνταξη αυτού του ψηφίσματος και θα λάβετε γνώση αυτού το συντομότερο δυνατό. Ευχαριστώ πολύ. Λήξη συνεδρία.